Συνάδελφοι, θέλω να αρχίσουμε, είναι η θέλησή μου αυτή. Καλώς σας καλωσορίζω. Αρχίζουμε με την έγκριση της ημερήσιας διάταξης που έχει διανεμηθεί <clears throat> από τις 26 Νοεμβρίου. Προτείνω δύο αλλαγές. Η μία, το πότε <clears throat> θα σας κάνω την ανακοίνωση των Προέδρων μετά τη συνάντηση των συντονιστών που θα γίνει στις 3 για να μην κάνουμε δύο ανακοινώσεις <clears throat> της Προεδρίας και καθυστερούμε. Δεύτερον, η ήττα συνεδρίαση, δηλαδή η παρουσίαση από τις σχετικές υπηρεσίες του Κοινοβουλίου της ενίας του e-meeting που λένε αλλά αργότερα και αυτό για να είναι περισσότεροι παρόντες και να μην το χάσουν. Αν δεν υπάρχει κανένα άλλο σχόλιο για την ημερήσια διάταξη, τότε λέω να την εγκρίνουμε. Θέλω να την εγκρίνουμε. Και περνάμε στο επόμενο σημείο. Η ακρόαση για τη μεταρρύθμιση του Ευρωπαϊκού Εκλογικού Νόμου. This hearing, uh, we are... Στην ακρόαση αυτή θα ασχοληθούμε και με την προετοιμασία νομοθέτικων ε, ρυθμίσεων της Επιτρόπης μας για την αλλαγή του εκλογικού νόμου της Ευρώπαικη Ένωσης. Ό, ίσως να θυμάστε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πάντοτε ήταν στο προσκήνιο και ζητούσε ενοποίηση του εκλογικού νόμου στις χώρες μέλη. Το 1998 είχε γίνει μια σοβαρή έκθεση που μιλούσε για την The member states ε? όχι αναλογικό για την αναλογικότητα για την, και για τη δημιουργία εθνικών και υπερεθνικών ψηφοδελτίων. Ο Ανδρέας Ντάφτιν είχε γράψει και είναι σήμερα ένας από τους εμπειρογνώμονές μας. Το 12, τον Ιανουάριο του 12, είχαμε πει ότι δεν υπήρχε ακόμη λόγος να προχωρήσουμε περισσότερο και να πάμε στην Ολομέλεια. Και γι' αυτό μετά τις ευρωπαϊκές εκλογές που βασίστηκαν σε εθνικούς εκλογικούς νόμους θα δούμε τι σήμαινε αυτό και το θέμα της αναλογικής εκπροσώπησης του συστήματος DONT για τη χορήγηση εδρών με ανοιχτά κλειστά ψηφοδέλτια και υπάρχουν και άλλα θέματα για θέματα όπως οι προεκλογικές δαπάνες κλπ. Και γι' αυτό θέλουμε να ξανασυζητήσουμε το θεμητό ερώτημα της ενοποίησης ή περισσότερης ενοποίησης του εκλογικού νόμου. Γι' αυτό κάνουμε την ακρόαση αυτή. Θα παρουσιάσω τους ομιλητές αργότερα, αργότερα. Αρχίζουμε όμως από τα σχόλια ενός άλλου ευρωπαϊκού οργάνου που ασχολείται και αυτό με το σημαντικό αυτό θέμα, τον κύριο Πολ Νέμιτ που είναι διευθυντής για τα βασικά δικαιώματα, τα θεμελιώδη στη Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης της Κομισιόν. Ορίστε κύριε Διευθυντά μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και να με συγχωρείτε για την αλλαγή στην ημερήσια διάταξη. Σας ευχαριστώ και για τη δυνατότητα που μου δίνετε να πω κάποια λόγια. Ευχαριστώ για το ότι ξεκίνησε η δουλειά τόσο σύντομα μετά τις εκλογές, γιατί όπως ξέρετε η μετεκλογική περίοδος είναι και προεκλογική και οπωσδήποτε η συμμετοχή στις εκλογές δεν είναι κάτι το οποίο αποφασίζεται τη μέρα των εκλογών. Τι εννοώ με αυτό. Μετράει βεβαίως ε, και η ημερομηνία των εκλογών όταν μιλάμε για τα ποσοστά της προσέλευσης. Αλλά το θέμα της συμμετοχής στη δημοκρατία δεν αποφασίζεται μόνο την ημέρα των εκλογών, αλλά χρειάζεται μια ευρύτερη προσέγγιση και βεβαίως ε, η εμπλοκή στη δημοκρατία δεν είναι μόνο η ψήφος, αλλά και η συμμετοχή στην πολιτική ζωή πριν και μετά τις εκλογές. Οπότε, όταν μιλάμε για συμμετοχή στις εκλογές, ε, είναι ένα ευρύτερο ζήτημα. Πρώτα απ' όλα το θέμα του πώς βλέπει ο κόσμος στην Ευρώπη, αλλά και το πώς εμπλέκεται γενικότερα στην δημοκρατία. Και εδώ πέρα θα ήθελα να αναφερθώ στα νούμερα που είχαμε δει στην προηγούμενη έκθεση για τη συμμετοχή στις ε, δημοτικές ε, και περιφερειακές εκλογές των Ευρωπαίων πολιτών. Βλέπουμε πως το πρόβλημα του ότι δεν συμμετέχουν αρκετοί στις εκλογές δεν περιορίζεται ή δεν αφορά ειδικά τις ευρωεκλογέ. Υπάρχει μία τάση γενικά του ότι η δεν αφορα ειδικα τις ευρωεκλογες υπαρχει μια ταση γενικα του οτι η προσελευση σε δευτερεύουσα σημασία εκλογές που δεν είναι δηλαδή εθνικές εκλογές είναι χαμηλή και σε δημοτικές περιφερειακές και στις ευρωεκλογές και βεβαίως πέρα από αυτό βλέπουμε και ότι πέφτουν και, πέφτει και ο αριθμός των μελών των πολιτικών κομμάτων και άλλες μορφές συμμετοχής. Σημαντικό λοιπόν είναι όταν μιλάμε για την συμμετοχή και τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας να το βλέπουμε στο ευρύτερο πλαίσιο του ότι πρέπει να λειτουργεί η δημοκρατία σε όλα τα επίπεδα γιατί συμφωνούμε με αυτή την πρόκληση ε, και είναι πράγματι κοινή αυτή η πρόκληση με κοινή και στις ε, δημοτικές ε, και περιφερειακές εκλογές από το, και πριν από το 1979 και μετά βέβαιως ήταν ζήτημα αυτό και τώρα για πρώτη φορά βλέπουμε πως υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ του αποτελέσματος των εκλογών και ε, του προτινόμενου Προέδρου της Κομισιόν. Αυτό μετά από συζήτηση και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά ε, και στον πανεπιστημιακό χώρο. Εγώ το 1998 ε, είχα ήδη δημοσιεύσει ένα άρθρο για την ε, έμεση εκλογή του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κάτι το οποίο με χαροποίησε ιδιαίτερα και έχω κορνιζάρει την σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 2013 όπου το σώμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συνέστησε πως ε, οι πολιτικές οικογένειες θα πρέπει να ορίσουν ένα κοινό υποψήφιο για πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Συνεισφέραμε λοιπόν και εμείς σε αυτό. Και στη σύσταση αυτή μάλιστα η Κομισιόν ζήτησε να εκμεταλλευτούμε την ε, συνθήκη της Λισαβόνας και να προτείνουμε υποψηφίους ε, μετά από τα αποτελέσματα των ευρωπαϊκών εκλογών, ζητάει από τα κόμματα να πούν ποιους θα στηρίξουν, ε, τα ευρωπαϊκά και τα εθνικά κόμματα. Και τα εθνικά κόμματα βεβαίως ε, να φροντίσουν να δείξουν σε ποια ευρωπαϊκή πολιτική οικογένεια ανήκουν. Τώρα συντάσσουμε μια έκθεση που αξιολογεί ακριβώς τον αντίκτυπο αυτών των στάσεων της Κομισιόν στις ε, ευρωεκλογέ του 2014 και ελπίζουμε να μπορέσουμε να την παρουσιάσουμε το πρώτο εξάμεινο του 2015 και αναμένουμε και τη συνεργασία μαζί σας γιατί θέλουμε η έκθεση αυτή να είναι μια έκθεση η οποία δεν θα αφορά απλώς ε, τα στατιστικά στοιχεία αλλά θα περιέχει και τις λοιπές δραστηριότητες, τα κοινωνικά μέσα, τα ευρήματα των κοινωνικών επιστημών για το πώς αντιλαμβάνονται οι πολίτες, ε, το γιατί ακριβώς ψηφίζουν, να μην κοιτά μόνο τους αριθμούς ε, της συμμετοχής. Όμως είναι σαφές πως η καινοτομία αυτή των εκλογών έχει την δυνατότητα να επιφέρει ε, ακόμη περισσότερη δημοκρατική νομοποίηση... στην ε, ευρωπαϊκή διαδικασία λήψης αποφάσεων, ένα σημαντικό βήμα στο να γίνει πιο δημοκρατική η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της. Και το ότι αυτή η Επιτροπή έχει δεσμευτεί να επιφέρει ακόμα πιο δημοκρατικές αλλαγές σημαίνει πως θα πρέπει να βρούμε κάποιους τρόπους για να εδρεώσουμε την ευρωπαϊκή διάσταση των ευρωεκλογών και να προωθήσουμε την δημοκρατική νομοποίηση. Σκοπεύουμε λοιπόν να κάνουμε ένα διάλογο με όλους τους ενδιαφερόμενους για να δούμε πώς θα εκμεταλλευτούμε καλύτερα το ποιοτικό στοιχείο των ευρωεκλογών του 2014, πώς θα το αναλύσουμε. Εδώ πέρα χρειαζόμαστε βεβαίως και τους πανεπιστημιακούς που βρίσκονται εδώ σήμερα και πρέπει να έχουμε μια περισσότερο ποιοτική ανάλυση ναι, όσον αφορά το μοντέλο αυτό των κορυφαίων κομματικών υποψηφίων. Και πρέπει επίσης να, για να έχουμε αυξημένη συμμετοχή, να δούμε τι θα γίνει. Γιατί σχεδόν σταμάτησε η πτωτική πορεία της ε, συμμετοχής. Έπεσε η συμμετοχή κατά μόλις 0,55% σε σχέση με 2% της προηγούμενης εκλογής και 4% στις προπροηγούμενες. Ο Τζο Βάιλερ, καθηγητής Ευρωπαϊκού Δικαίου και τώρα πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου στη Φλωρεντία, το 1979 δημοσίευσε ένα βιβλίο στο οποίο προέβλεψε πως η συμμετοχή στις ευρωεκλογές θα αυξηθεί παράλληλα με τις αυξημένες αρμοδιότητες του Κοινοβουλίου, δηλαδή με την αύξηση της συναπόφασης. Και ο ίδιος ο Τζοβάιλερ πριν από ένα χρόνο περίπου είπε πως λυπόταν για το ότι έκανε λάθος στην πρόβλεψή του αυτή. Είδαμε αύξηση της ε, συμμετοχής του Κοινοβουλίου όσον αφορά τη συναπόφαση για το δημοκρατικό έλεγχο και τη λήψη αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μείωση της συμμετοχής στις ευρωεκλογές. Οπότε, απλώς το να λέμε ότι με μεγαλύτερη σημασία του ερετού σώματος θα έχουμε περισσότερο ενδιαφέρον των πολιτών, δεν αποδείχτηκε σωστό. Πέρα από το την λοιπόν υπάρχει και το ζήτημα της επικοινωνίας και πρέπει να κινητοποιήσουμε τον κόσμο όλοι για να μπορέσουμε ακριβώς ε, να πλαισιώσουμε τις αυξημένες αρμοδιότητες του Κοινοβουλίου με αυξημένη συμμετοχή στις ευρωεκλογέ. Περισσότερα μπορούν και πρέπει να γίνουν και εγκαίρως όχι μόνο λίγο πριν τις εκλογές για να μπορέσουμε να ενημερώσουμε τους ε, πολίτες και το πώς ε, οι ευρωεκλογέ επηρεάζουν την ζωή τους. Ταυτόχρονα θα προσπαθήσουμε να διαφυλάξουμε τα πολιτικά δικαιώματα των ε, Ευρωπαίων πολιτών που μετακινούνται. Το δικαίωμα των Ευρωπαίων πολιτών να ψηφίζουν και να είναι υποψήφιοι στις ευρωεκλογές στο κράτος μέλος όπου κατοικούν με τις ίδιες συνθήκες με τους υπηκόους αυτού του κράτους μέλους είναι βασικό δικαίωμα του Ευρωπαίου πολίτη στο άρθρο 22 και στο άρθρο 39 στο άρθρο 22 της συνθήκης και στο άρθρο 39 της Χάρτας των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και αναφέρεται και στην Οδηγία 9309. Θα ήθελα εδώ πέρα να τονίσω πως σκοπεύουμε να απλοποιήσουμε τη διαδικασία για να κατεβαίνουν υποψήφοι οι ε, Ευρωπαίοι πολίτες που είναι σε άλλο κράτος μέλος ε, από το δικό τους. Σύμφωνα με τις ε, οδηγίες, σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 20 του 2001 δεν πρέπει να προσκομίσουν κάποιο πιστοποιητικό ότι δεν έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα, απλά υπογράφουν μια βεβαίωση την οποία μετά ελέγχει το αρμόδιο κράτος μέλος. Από ό,τι φαίνεται υπήρχε αύξηση των πολιτών της Ένωσης που ζουν σε άλλο κράτος μέλος ε, και κατέβηκαν υποψήφοι από 81, κατεβήκαμε σε 150, ανεβήκαμε σε 152 το 2014. Επίσης, σκοπεύουμε να αυξήσουμε την ενημέρωση των πολιτών και να φέρουμε την ευρωπαϊκή πολιτική διαδικασία πιο κοντά στον πολίτη. Σύμφωνα λοιπόν με την ε, διαδικασία για τα δικαιώματα και την ε, υπηκότητα των ε, πολιτών. Σκοπεύουμε να φέρουμε την πολιτική ζωή της Ευρωπαϊκής Ένωσης πιο κοντά στον πολίτη και να πω εδώ πέρα για τους καθηγητές που είναι παρόντες πως μέχρι τον Φεβρουάριο του 2015 είναι η προθεσμία για υποβολές προσφορών, ε, προτάσεων, τις οποίες ε, θα χρηματοδοτήσουμε. Όσον αφορά τώρα το πώς ε, εφαρμόζονται αυτοί οι κανόνες από τα κρατημέλη και πώς εφαρμόστηκαν στις ευρωεκλογές του 2014, θα προσπαθήσουμε να χρησιμοποιήσουμε το νέο κεκτημένο για να διευκολύνουμε τη δημοκρατική συμμετοχή των πολιτών της Ένωσης. Η συζήτηση που ξεκινάει σήμερα για την πιθανή ανάγκη μεταρρύθμισης της νομοθεσίας του 1976 και των κοινών αρχών εκλογής των ευρωβουλευτών μας δίνει την δυνατότητα να ξανασκεφτούμε αυτά τα ζητήματα μετά τις τελευταίες εκλογές. Τα κρατημέλη, τα κόμματα, think tanks και πανεπιστημιακοί έχουν προσκληθεί επίσης να συνεισφέρουν σε αυτή τη διαδικασία ο καθένας από τη σκοπιά του. Κατά τον τρόπο αυτό θα μπορέσουμε να ενισχύσουμε περαιτέρω την ευρωπαϊκή διάσταση των επόμενων εκλογών και την ε, εμπλοκή των ψηφοφόρων και να αυξηθεί η δημοκρατική νομιμοποίηση της λήψης αποφάσεων. Και βεβαίως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεργαστεί μαζί σας πλήρως. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι είναι καλά νέα για μας ε, κύριε Νέμιτς και χαίρομαι που θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε. Και αυτή τη φορά ελπίζω να τα καταφέρουμε και να φτάσουμε και μέχρι την Ολομέλεια. Να περάσουμε τώρα στην ακρόαση. Αυτή καθε αυτή και να ακούσουμε πρώτα δύο εμπειρογνώμονες. Πρώτα θα λάβει το λόγο ο Άντριου Νταφ. Δεν ξέρω αν χρειάζεται συστάσεις. Ήταν χρόνια εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ανήκει στην οικογένεια των φιλελεύθερων και δημοκρατών. Και φυσικά ήταν και εισηγητής σε σειρά εκθέσεων που σχετίζονται με το θέμα που συζητούμε σήμερα. Άντριου λοιπόν έχει το λόγο. Um, uh, uh, Κυρία Πρόεδρε, Ντανούτα, καταρχάς να σε ευχαριστήσω που με προσκάλεσες να μιλήσω εδώ. Είναι μεγάλο προνόμιο νομίζω για πρώην Ευρωβουλευτή να καλείται να εξηγηθεί. Και μάλιστα επειδή η Επιτροπή και εγώ κάναμε προσπάθειες για τη μεταρρύθμιση της εκλογικής διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αυτές οι προσπάθειες απέτυχαν και σε κάποιο βαθμό όλοι αναλαμβάνουμε ε, ευθύνες για αυτή τη σχετική αποτυχία. Αλλά Από τότε που έχασα την έδρα μου το Μάιο, μπόρεσα να σκεφτώ λίγο περισσότερο και να διαβάσω πολλά περισσότερα για ένα θέμα το οποίο θεωρώ ότι είναι μια βαθύτερη κρίση της ευρωπαϊκής δημοκρατίας. Δεν είναι κάτι το οποίο ορίζεται με στενά όρια ως απλώς ε, η εκλογική διαδικασία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Νομίζω ότι το αποτέλεσμα της ε, χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης εν μέρη ενέτεινε τις φυγόκεντρες πιέσεις ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω ότι δεν υπάρχει καμία χώρα που αυτή τη στιγμή δεν αντιμετωπίζει σοβαρά εσωτερικά και συνταγματικά προβλήματα και αναταραχές. Και φυσικά δεν μπορεί κανείς να αποκλείσει και το δεχόμενο της ε, ίδιας της διάλυσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει θέμα δημοκρατικής νομιμοποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εν μέρη προκύπτει και από τους ίδιους τους πολίτες που δεν ε, προσέχουν αρκετά. Εν μέρη είναι ευθύνη των Εθνικών Κοινοβουλίων και των Εθνικών Πολιτικών Κομμάτων που σχεδόν έχουν παραιτηθεί και δεν υποστηρίζουν και δεν προωθούν το ευρωπαϊκό όραμα λόγω άγνοιας ή και φθόρνου κάποιες φορές ή και τα δύο μαζί. Και εν μέρη είναι και ευθύνη των ίδιων των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων που ακόμα προσπαθούν να αντιληφθούν πώς λειτουργεί ένα σύστημα διακυβέρνησης το οποίο είναι περίπλοκο ε, και αρκετά δύσκολο και αδιάφανο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει πάρα πολύ σημαντικές εξουσίες ε, μέσω του δικαιώματος πρωτοβουλίας. Υπάρχει καταρχάς το άρθρο 2.23 ε, της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ε, προσπάθεια ε, ενιαίας εκλογικής διαδικασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και υπάρχει και το άρθρο 14 σημείο 2 της ε, ε, νέας συνθήκης Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη Λισαβόνα και μετά που επιτρέπει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να προτείνει ένα σύστημα κατανομής ευρών μεταξύ των ε, κρατών μελών του Κοινοβουλίου. Θα ήθελα να επιμείνω σε αυτό. Δεν είναι απλώς δικαιώματα τα οποία απολαμβάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά και καθήκοντα, τα οποία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να εκπληρώσει. Και από προσωπική πείρα γνωρίζω ότι είναι μάλλον δύσκολο για το ίδιο το Κοινοβούλιο να αποδεχτεί μια μεταρρύθμιση μιας εκλογικής διαδικασίας όταν υπάρχουν τόσα συμφέροντα των ίδιων των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αφορούν και τη σταδιοδρομία τους και τις συντάξεις τους τα θέματα αυτά. Επομένως είναι πολύ πιο εύκολο να παραμείνει κάποιος στο status quo και είναι πολύ δύσκολο να το αλλάξει κανείς. Και αν η σημερινή σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θέλει να βελτιώσει τα πράγματα σε σχέση με τις προηγούμενες θητείες, όντως είναι κατάλληλη στιγμή να ξεκινήσουμε τώρα και να είμαστε έτοιμοι για το 2019. Καταρχάς, το θέμα των ε, ευρωπαϊκών ε, ψηφοδελτίων. Νομίζω ότι η ιδέα του speech and candidate, ε, του επικεφαλής των ψηφοδελτίων, είναι επιτυχής λύση και εξέπληξε αρκετούς, μεταξύ των οποίων και εμένα, διότι κατάφερε να σπάσει, αν θέλετε, αυτό το καλούπι το οποίο ε, επικρατούσε στις προηγούμενες επιλογές, ε, υπήρχαν και πάρα πολλές διαφιλονικίες επ' αυτού και κυρίως η ίδια η πολιτική τάξη, η ελίτ της Ευρώπης δεν ήθελε να δεχτεί. Επειδή όμως ακριβώς ε, ήταν επίμαχο ζήτημα, εξέπλησε και τους Πρωθυπουργού και τους προέδρους και γι' αυτό ακριβώς ε, είναι μια αρχή μόνο και θα πρέπει να βελτιωθεί περαιτέρω και να αναθεωρηθεί. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφώνησε ότι θα πρέπει να ξαναδεί το σύστημα για το διάδοχο του Πρόεδρου Γιούνκερ και θα ήθελα να ε, συστήσω στο Κοινοβούλιο να αναλάβει πρωτοβουλία από αυτού ώστε τουλάχιστον να προσπαθήσει να διασώσει την ουσία του όλου αυτού πειράματος ε, για το 2014 για τον επικεφαλής της λίστας και το πείραμα αυτό να καταλήξει σε ένα λογικό συμπέρασμα που θα είναι η ε, πρώτη των ψηφοδελτίων να μπουν σε ένα υπερεθνικό ψηφοδέλτιο μέσω του οποίου θα εκλέγονται τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για μια πανευρωπαϊκή επικράτεια. Αν φυσικά γίνει αυτό, καταρχάς θα συμπεριλαμβάνεται εκεί και ο υποψήφιος πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Αλλά επίσης δεν θα υπάρχει και πρόβλημα με το συνταγματικό δικαστήριο της Γερμανίας διότι εκεί γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχει ομοιομορφία. Θα υπάρχει μια ευρωπαϊκή διάσταση στις ευρωεκλογέ πλέον, αν υπάρχει ευρωπαϊκό ψηφοδέλτιο και τα πολιτικά κόμματα θα γίνουν πραγματικά ε, κόμματα τα οποία θα κάνουν κανονική προεκλογική εκστρατεία. Και θα αποτελέσει φυσικά αυτό και ένα δώρο για το εκλογικό σώμα, διότι δεν θα χρειάζεται να ρίξει μόνο μία ψήφο για τους περιφερειακούς ή τους εθνικούς ευρωβουλευτούς τους, αλλά θα ψηφίσει και μία δεύτερη φορά για έναν Ευρωπαίο Ευρωβουλευτή. Αν το καταφέρουμε αυτό, και στο παράρτημα 3 της μελέτης μου, παρουσιάζω και με απλήρη αναθεώρηση της πράξης του 1976. Αν λοιπόν καταφέρουμε να έχουμε αυτή τη λύση θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε και άλλα πράγματα. Θα μπορούσαμε ίσως να έχουμε και ένα όριο για την ε, ηλικία των υποψηφίων. Να σκεφτούμε και θέματα φύλου. Να εξετάσουμε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των ανοιχτών και κλειστών ψηφοδελτίων. Το να σκεφτούμε και το να έχουμε ε, συγκεντρωτικά ημέρες ε, ψηφοφορίας και να υπάρχουν και συγκεκριμένα δικαιώματα για τους ευρωβουλευτές, να πληρώσουμε τυχόν κενά και να καθορίσουμε και μία εκλογική αρχή σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το οποίο, η οποία θα είναι υπόλογη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο Κοινοβούλιο. Σε αυτό το πλαίσιο μπορούμε να βελτιώσουμε και το καθεστώς των πολιτικών κομμάτων που παρά τις ε, πολύ μεγάλες μάχες που δόθηκαν στο προηγούμενο κοινοβούλιο, πραγματικά χρειάζεται ουσιαστικές βελτιώσεις. Εδώ μπορούμε να διευρύνουμε και το δικαίωμα του εκλέγην και φυσικά να ρυθμίσουμε και θέματα ε, συγκέντρωσης ε, στατιστικών στοιχείων ε, για το πληθυσμό. Αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα, το οποίο θεωρώ ότι θα πρέπει να απασχολεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το δεύτερο αφορά την κατανομή των εδρών. Και εδώ προσφάτως διαπιστώσαμε ότι ακόμα και οι 11 έδρες της Κροατίας δημιούργησαν έρηδες και εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο αλλά και μεταξύ Συμβουλίου Και είναι εξαιρετικά καλό το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφώνησε το 2013 να υπάρχει ένας συγκεκριμένο τύπος υπολογισμού ο οποίος θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί εγκαίρως για τις εκλογές του 2019. Υπάρχουν εργασίες ε, του καθηγητή Πούκελσχάιμερ και του υποφαινόμενου ε, ένα πρόγραμμα το οποίο αποκαλούμε CAMCOM είναι ο συμβιβασμός του Cambridge το οποίο συνεψίζω στη μελέτη μου ένα σύστημα το οποίο θα ήταν αποτελεσματικό αν υπήρχαν επιπλέον 25 υπερεθνικές έδρα των 751 ευρών και υπολογίζει και ε, τι θα μπορούσε να γίνει στην περίπτωση που αυτές οι 25 αφαιρεθούν από τις 751. Εάν ε, έχουμε μία συνολική, δίκαιη και ε, μια λύση που αντιμετωπίζει τις επικρίσεις ε, του γερμανικού, του γερμανικού συνταγματικού δικαστηρίου και καταφέρουμε να βρούμε μια τέτοια λύση για τον υπολογισμό της κατανομής των ευρών, και θα πρέπει να φροντίσουμε να μην υπάρχει παραβίαση ε, των συνθήκων και της νομοθεσίας. Το παράρτημα της ε, μελέτης μου έχω προτείνει μία διαδικασία δύο σταδίων για αυτό το ΚΑΝΚΟΝ. Η πρώτη θα εφαρμοστεί το 2019. Αν αλλάξει όμως η κατανομή των ισορροπιών μεταξύ των κρατών μελών στο Κοινοβούλιο, τότε θα πρέπει να δούμε και τι γίνεται με την ισορροπία ε, εξουσιών στο Συμβούλιο. Θα πρέπει να τονίσουμε εδώ ότι στην πραγματικότητα είμαστε ένα νομοθετικό σώμα με δύο βουλές. Και η δεύτερη βουλή θα πρέπει να επανεξεταστεί και να ρίξει μια νέα ματιά στο εκλογικό σύστημα. Είναι αλήθεια ότι η μεταρρύθμιση της κατανομής των εδρών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα τιμωρήσει, αν θέλετε, τις χώρες μεσαίου μεγέθους, οι οποίες αυτή τη στιγμή εκπροσωπούνται περισσότερο από όσο θα έπρεπε. Το σωστό λοιπόν και το δίκαιο θα ήταν η αντιστάθμιση για τις ε, απώλειες των εδρών των μεσαίου μεγέθους χωρών μέσω αύξησης της ε, ισχύου τους ε, στο Συμβούλιο. Και υπάρχει ένας μαθηματικός τύπος που βασίζεται στην τετραγωνική ρίζα και δίνει στα κράτη ε, μία στάθμιση ε, αντιστρόφως ανάλογη του μεγέθους τους. Υπήρχε ε, για πολύ σύντομο διάστημα περαστική στη συνταγματική συνθήκη, αλλά νομίζω ότι πρέπει να την ξαναλάβουμε υπόψη αυτή τη λύση. Τρία στοιχεία. Το υπερεθνικό ψηφοδέλτιο, η κατανομή των εδρών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η αναθεώρηση των βαρών στο Συμβούλιο αποτελούν μια δέσμη μέτρων τα οποία θα μας οδηγήσουν σε μια βιώσιμη δημοκρατική επίλυση αυτών των ευαίσθητων θεμάτων. Τέλος, να πω δύο λόγια για τη διαδικασία, η οποία θα πρέπει να είναι ε, εξίσου νομιμοποιημένη με το αποτέλεσμα. Και εδώ γνωρίζουμε ότι θα υπάρξει μια συνταγματική συνέλευση. Δεν ξέρουμε πότε θα γίνει, αλλά η πεποίθησή μου ότι μάλλον θα γίνει ε, αρκετά σύντομα και δεν θα καθυστερήσει πολύ και θα πρέπει να αντιμετωπίσει κυρίως το θέμα της ε, Δημοσιονομικής Ένωσης. και της μεταρρύθμισης του χρηματοπιστωτικού συστήματος Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να διορθώσει κάποια από τα πιο αδύναμα στοιχεία της ε, συνθήκης της Λισαβόνας, να εξυγχρονίσει κάποιες ε, παροχημένες κοινέ πολιτικές και να αντιμετωπίσει και το βρετανικό ζήτημα. Μέσα λοιπόν σε αυτή τη δέσμη μέτρων πρέπει η μεταρρύθμιση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να συμπεριληφθεί και να συγχαρώ την Επιτροπή σας που ξεκινά ε, ε, τόσο νωρίς και μάλιστα με ιδιαίτερο θάρρος για αυτή τη τόσο σημαντική κίνηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Άντριου και για τα ενθαρρυντικά σου λόγια και για τα απόψεις σου και να περάσουμε τώρα στον καθηγητή Πούκελσχάιμεν, ο οποίος είναι από το Πανεπιστήμιο του Άουσμπουργκ, ε, του Τμήματος των Μαθηματικών και νομίζω ότι είναι και πολύ δραστήριος στο London School of Economics στο Λονδίνο. Θα ήθελα να ακούσω λοιπόν και τη δική σας την άποψη επί του ζητήματος και κατόπιν θα γίνει μια συζήτηση ε, και για τις δύο παρουσιάσεις. Κύρια Πρόεδρε, Κύριε... Αγαπητοί κύριοι βουλευτές, σας ευχαριστώ που με καλέσατε στην συνεδρίαση αυτή για το θέμα της ε, νομοθεσίας των ευρωεκλογών. Η πρόοδος ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ήταν εντυπωσιακή και έχει γίνει πλέον ένας πυλώνας της δημοκρατικής δομής της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και οι ευρωβουλευτές εκλέγονται με άμεση καθολική ψηφοφορία από τους Ευρωπαίους πολίτες. Εγώ θα έλεγα πως ε, το ποτήρι είναι μισογεμάτο. Εμείς έχουμε χωρίσει την έκθεσή μας σε κομμάτια α, β και γ. Κοιτάμε τις επιχειρησιακές πτυχές και το εάν ε, συμμορφώνονται οι διαδικασίες αυτές με τους πολιτικούς στόχους. Ως πηγές είχαμε τα παλαιότερα έγγραφα της Επιτροπής σας και του Κοινοβουλίου, επίσης ε, την ε, σχετική βιβλιογραφία, αν και επειδή αυτή είναι πολύ εκτεταμένη βεβαίως, έπρεπε να γίνουν κάποιες επιλογές και βασιστήκαμε και στην δικιά μας τη δουλειά, την μαθηματική ανάλυση εκλογικών συστημάτων, Οπότε θα ξεκινήσω με το πρώτο μέρος. Ποιο είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι πως το εκλογικό σώμα κατευθύνεται λάθος. Το μεγαλύτερο ελάττωμα του τωρινού εκλογικού συστήματος είναι πως κατευθύνει λάθος το εκλογικό σώμα. Η εκστρατεία εστιάζεται σε ηγέτες που διαμορφώνουν την πολιτική σκηνή εντός του κράτους μέλους, αλλά δεν ανταγωνίζονται για κάποιες έδρες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι ψηφοφόροι παίρνουν ψηφοδέλτια με κόμματα εθνικά του κάθε κράτους μέλους, τα οποία όμως είναι αόρατα ουσιαστικά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τα 160 περίπου εθνικά κόμματα που παρουσιάζονται στο Ευρωπαϊκό Εκλογικό Σώμα τελικά καταλήγουν σε μια χούφτα πολιτικών ομάδων, οι οποίες όμως δεν εμφανίζονται ενώπιον του εκλογικού σώματος. Για να αναφέρω λοιπόν μία μονοπήγη, υπάρχει αναντιστοιχία μεταξύ του θεσμικού ρόλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εντός της Ένωσης και της διάκρισης των εξουσιών της και του επίπεδου κομματικού ανταγωνισμού των ευρωεκλογών. Οπότε, εάν το Ευρωκοινοβούλιο θέλει περισσότερη ομοιομορφία στον εκλογικό νόμο, τότε απαραίτητο προαπαιτούμενο είναι η σύσταση ευρωπαϊκών κομμάτων για να παίξουν τον σωστό ρόλο στις ευρωεκλογέ. Αυτή είναι η άποψή μας. Υπάρχει πολύ σχετική βιβλιογραφία από πολιτικούς επιστήμονες, συνταγματολόγους και πολιτικούς. Εμείς βεβαίως είμαστε μαθηματικοί, δεν μπορούμε να σχολιάσουμε το πώς θα δημιουργηθεί ένα πανευρωπαϊκό σύστημα κομμάτων. Ε, ανταυτού υποθέτουμε πως θα υπάρχουν τέτοια κόμματα και θα κατεβαίνουν στις εκλογές. Ξεκινώντας με αυτή την υπόθεση, προτείνουμε ένα σύστημα μετάφρασης των ψήφων σε έδρες, το οποίο ταιριάζει με το συναγματικό πλαίσιο της διπλής αναλογικότητας. Πριν συνεχίσουμε να κάνουμε μια παρέκβαση για να εξηγήσουμε τι εννοούμε πανευρωπαϊκά κόμματα εδώ πέρα. Είναι λιγότερο περιοριστικό από τον όρο πολιτικά κόμματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο που περιέχεται στον κανονισμό χρηματοδότησης. Εμείς θεωρούμε πως το Πανευρωπαϊκό Κόμμα είναι ένας πολιτικός οργανισμός που στο πρόγραμμά του και στις δραστηριότητες του ε, τηρεί τις αρχές πάνω στις οποίες ιδρύθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση και ε, συμμετέχει ή σκοπεύει να λάβει μέρος στις ευρωεκλογές. Αυτά απαιτούμε εμείς. Στις περισσότερες περιπτώσεις ένα τέτοιο κόμμα θα δραστηριοποιείται σε δύο ή περισσότερα κράτη-μέλη, ίσως και σε όλα, όμως ο ορισμός δέχεται, ε, πώς μπορεί το ακόμα να βρίσκεται μόνο και σε ένα κράτος μέλος. Γιατί το σύστημα θα πρέπει να δέχεται και νέα κόμματα, τα οποία βεβαίως δεν μπορεί παρά να ξεκινήσουν από χαμηλά. Δεύτερον, ποια είναι η λύση. Η λύση λέγεται διπλή αναλογικότητα, η οποία κατανέμει τις έδρες ε, με δύο κριτήρια. Πρώτον, το πώς ε, κατανέμεται το εκλογικό σώμα στα διαφορά κόμματα και δεύτερον, πώς χωρίζεται σε ε, εδαφικές περιφέρειες. Τι μορφή έχει δηλαδή η διπλή αναλογικότητα όταν εφαρμόζεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η πολιτική διατάσταση ε, βεβαίως είναι το πώς πηγαίνουν τα κόμματα. Η εδαφική διάσταση είναι η κατανομή των εδρών στα κράτη-μέλη της Ένωσης ή όπως τα λέει η συνθήκη ε, αφορά την σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η διπλή αναλογικότητα θα ισχύει ανεξαρτήτως του, της ε, σύνθεσης είτε αυτή θα είναι αποτέλεσμα διαπραγμάτευσης όπως το παρελθόν είτε μέσω μιας μόνιμης και διαφανούς λύσης. Η διπλή αναλογικότητα απαιτεί ε, ένα υποσύνολο το οποίο θα είναι ένα υποσύνολο εδρών το οποίο θα είναι προκαθορισμένο ανά κράτος μέλος και έχουμε δύο βήματα μία υπερκατανομή και μία υποκατανομή. Η υπερκατανομή αντικατοπτρίζει τα πανευρωπαϊκά αποτελέσματα. Όλες οι διαθέσιμες έδρες κατανέμονται ανάλογα με το σύνολο των ψήφων των πανευρωπαϊκών κομμάτων. Βλέπουμε εδώ πέρα ένα δείγμα υπερκατανομής στον πίνακα 1 των εντύπων που σας έχουμε δώσει. Είχαμε δηλαδή τα αποτελέσματα των ε, προηγούμενων ευρωεκλογών του 2009. Επειδή δεν υπήρχαν τέτοια κόμματα το 2009, τα αντικαταστήσαμε με τις πολιτικές ομάδες που σχηματίστηκαν στην αρχή της τότε θητείας. Το σύνολο των ψήφων θεωρούμε πως είναι το σύνολο των ψήφων που συγκέντρωσαν τα εθνικά κόμματα που μπήκαν σε αυτή την ομάδα. Και έχουμε και τους μη εγγεγραμμένους ως μια ψεύδο ομάδα θα έλεγα. Οπότε ο πίνακας συμπεριλαμβάνει και 144 εκατομμύρια ψήφους που τελικά έκριναν τις ε, ευρωεκλογές εκείνες. Η υπερκατανομή στον πίνακα 1 αντιμετωπίζει ε, με ίσο τρόπο όλες τις ψήφους ανεξαρτήτως ε, κράτους μέλους. Κάθε 120.000 ε, ψήφου, ψήφοι αντι, αντιστοιχούν σε μία έδρα. Και έτσι υπάρχει εκλογική ισότητα μεταξύ όλων των πολιτών της Ένωσης όταν μιλάμε για τις πολιτικές προτιμήσεις. Αυτή τη στιγμή η εκλογική ισότητα δεν υπάρχει στο πρωτογενές δίκαιο της Ένωσης. Από την άλλη, οι συνθήκες ε, είναι γεμάτες υποσχέσεις για ισότητα μεταξύ των πολιτών της Ένωσης και όλα τα κράτη-μέλη θεωρούν πως η εκλογική ισότητα είναι μία από τις πέντε αρχές της ε, εκλογικής κληρονομιάς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η ΕΣΔΑ, την οποία έχει υπογράψει η Ένωση, επίσης ε, αποδίδει μεγάλη σημασία στην εκλογική ισότητα. Εμείς προτείνουμε η Ένωση να δώσει στους πολίτες ακριβώς την ε, ισότητα της ψήφου. Αυτό ζητάμε μόνο ως αλλαγή στην συνθήκη. Και καταλήγουμε μετά με μια υποκατανομή εδρών ανά κόμματα και κράτη-μέλη. Αυτό είναι κάπως πιο δύσκολο, καθώς πρέπει εδώ πέρα να υπάρχουν και να πληρούνται δύο όροι. Οι έδρες της υποκατανομής πρέπει να αντιστοιχούν και στα κόμματα και στα κράτη-μέλη. Ο πίνακα 2 μας δείχνει ένα δείγμα πάλι με βάση τις εκλογές του 2009. Τα, τα ονόματα των κομμάτων και ο αριθμός των εδρών τα έχουμε αντιγράψει από την υπερκατανομή. Η αριστερή στήλη μας δείχνει τα κράτη-μέλη και τις έδρες που έχουν. Οι έδρες αυτές ε, είναι ως αποτέλεσμα του αριθμού των ψήφων επί του ποσοστού του κράτους μέλους και του ποσοστού του κόμματος σε αυτό το κράτος μέλος. Μπορείτε λοιπόν να παρατηρήσετε εδώ πέρα ανά στήλη της έδρες και βεβαίως ε, ανά οριζόντια το ποσοστό και θεωρούν πως αυτή η διπλή αναλογικότητα ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες ε, της Ένωσης. Το θέμα είναι πώς θα φτάσουμε εκεί. Το βασικό εμπόδιο παραμένει βεβαίως η δημιουργία ενός συστήματος πανευρωπαϊκών κομμάτων, αλλά υπάρχουν και άλλα ζητήματα που πρέπει να μας απασχολήσουν όταν ε, μιλάμε για καταμέτρηση των ψήφων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Υπάρχουν διαφορετικά εκλογικά συστήματα στα 28 κράτη-μέλη. Η εναρμόνιση βεβαίως που απαιτείται έχει χαμηλό κόστος, όμως ψηφοδέλτια στην περίπτωση μίας ενιαίας ψήφου δημιουργούν κάποιο πρόβλημα καθώς δεν υπάρχει πλέον μια κάποια προσωποποίηση σε σχέση με τα κόμματα. Ένας ε, κοινό παρονομαστής ε, αναλογικά με το κάθε κράτος μέλος μπορεί να, πάει, να οδηγεί στην εισαγωγή ανοιχτών ληστών εκεί όπου αυτές δεν υπάρχουν. Αξίζει βεβαίως να το δούμε το ζήτημα, αλλά εδώ πέρα δεν το εξετάζουμε περαιτέρω. Επιπλέον, οποιοδήποτε επανασχεδιασμός θα πρέπει να προωθήσει την ηλεκτρονική ψηφοφορία που θα γίνει απαραίτητη σε μελλοντικέ εκλογές ε, δεδομένης ε, και της ε, κινητικότητας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέρος γάμα τώρα. Πώς θα φτάσουμε εκεί. Τρεις ενδιάμεσες ρυθμίσεις για το 2019. Η σύσταση πανευρωπαϊκών κομμάτων που θα κατεβαίνουν στις ευρωεκλογές ίσως χρειαστεί περισσότερο χρόνο από μια θητεία πεντετών. Δέκα χρόνια πρέπει να αρκούν. Οπότε προτείνουμε να ε, καθορίσουμε από τώρα την διπλή αναλογικότητα για να ξεκινήσει από το 2024. Και έτσι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ακολουθήσει το παράδειγμα άλλων κοινοβουλίων ε, που όταν κάνουν μεγάλες αλλαγές ε, αυτές δεν ισχύουν από την τωρινή θητεία αλλά από την επόμενη. Για τις επόμενες εκλογές του 2019 προτείνουμε τρεις ενδιάμεσες ρυθμίσεις ε, που θα ενθαρρύνουν τον σχηματισμό πανευρωπαϊκών κομμάτων. Οι τρεις προτάσεις μπορούν να ενσωματωθούν στην εκλογική νομοθεσία. Έχουμε πρώτα απ' όλα ένα ευρωπαϊκό ψηφοδέλτιο και ευρωπαϊκό εκλογικό μέτρο. Το τρίτο θέμα, οι ε, ή υπερεθνικές λίστες, ε, θα ισχύσει μόνο το 2009, καθώς θα περιτεύει όταν υιοθετηθεί η διπλή αναλογικότητα. Η πρώτη πρόταση είναι τα ψηφοδέλτια να έχουν το έμβλημα και όνομα του Πανευρωπαϊκού Κόμματος ε, στο οποίο ανήκει το Εθνικό Κόμμα πάνω από το έμβλημα και όνομα του Εθνικού Κόμματος. Πιθανώς τα υφιστάμενα, υφιστάμενες ε, κοινοβουλευτικές ομάδες να αποτελέσουν τον πυρήνα των ευρωπαϊκών κομμάτων. Οπότε τα εθνικά κόμματα ξέρουν ήδη τώρα σε ποιο ευρωπαϊκό κόμμα θα ανήκουν και μπορεί εύκολα να ακολουθήσουν αυτή την πρόταση. Τα κόμματα τα οποία δεν είναι συνδεδεμένα θα έχουν ένα κενό διάστημα πάνω από το δικό του σήμα ακριβώς για να φαίνεται ότι δεν έχουν κάποια ευρωπαϊκή προοπτική. Οπότε η πληροφορία πάνω στο ψηφοδέλτιο δεν θα είναι καθαρά εγχώρια. Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας υποθέτουμε ότι τα κόμματα θα διαφημίζουν τα ψωδελτιά τους και το νέο σχέδιο θα διαδοθεί και θα δώσει την αίσθηση μιας ευρωπαϊκής προοπτικής στους ψηφοφόρους και γενικότερα θα είναι ευκολότερο από ότι τώρα οι ψηφοφόροι να έχουν μια σαφή άποψη των ευρωπαϊκών επιλογών τους. Η δεύτερη πρόταση σκοπεύει βεβαίως να ανταμείψει τα κόμματα για την προσπάθειά τους να γίνουν ευρωπαϊκό κόμμα και να επεκταθούν σε πολλά κράτη-μέλη. Το σκεπτικό είναι να μειωθεί το ανώτατο 5% που ορίζει το άρθρο 3 του εκλογικού νόμου που α, αναλόγως με το πώς εξαπλώνονται τα κόμματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παραδείγματος χάρη, μπορεί να έχουμε την εξής μορφή εκλογικού ορίου σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση αρχίζουν να μετράν οι ψήφοι μόνο εάν το κόμμα συγκεντρώσει τουλάχιστον 5% των έγκυρων ψήφων σε ένα κράτος μέλος ή 4% των έγκυρων ψήφων σε δύο κράτη-μέλη ή 3% σε τέσσερα κράτη-μέλη ή 2% σε 8 κράτη-μέλη. Έτσι, ε, αυτό δεν θα ισχύει βεβαίως για ανεξάρτητους υποψηφίους και αυτό μπορεί να ρυθμιστεί μετά με εθνικές διατάξεις. Η τρίτη πρόταση προσφέρει στα πανευρωπαϊκά κόμματα συγκεκριμένη ανταμοιβή για να γίνουν ευρωπαϊκά κόμματα, δηλαδή έδρες που θα είναι πλέον αντικείμενο ε, ευρωπαϊκού ανταγωνισμού. Οι διεθνείς ε, λίστες αναφέρονται και στην έκθεση της Επιτροπής σας του 2011. Εξηγούμε αυτή την ιδέα και λέμε πως θα γίνει πλέον παροχημένη όταν ευρεωθεί η διπλή αναλογικότητα. Δεδομένη της μεταβατικής φύσης του μέτρου, η άπαξ εφαρμογή του το 2019 θα είναι συμβατή με το υφιστάμενο πρωτογενές δίκαιο. Έχουμε τώρα εδώ πέρα μια πρώτη προσέγγιση. Η δική μας η προσέγγιση εξαρτάται από το ότι η σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα είναι αποτέλεσμα μιας σταθερής ε, λύσης όπως παραδείγματος χάρη ο συμβιβασμός του Κέμπριτζ ή μια τέτοια παραλλαγή. Όταν κάνουμε αναγωγή στην τωρινή σύνθεση, σημαίνει πως 25-26 έδρες θα πρέπει να ανακατανεμηθούν. Οι περισσότερες από αυτές τις έδρες πηγαίνουν από μεσαία κρατημέλη σε μεγαλύτερα και λίγες σε μικρότερα. Προτείνουμε οι έδρες αυτές να μην πάνε στα κράτη αυτά, ανταυτού να μείνουν κατά μέρος για να κατανεμηθούν με βάση τα, α, τις υπερεθνικές λίστες, όπως αναφέρει η έκθεση του 2011. Εκ πρώτης όψεως φαίνεται πως ε, τα κράτη-μέλη ε, θα επωφεληθούν από τη μεταφορά αυτή όμως το βάρος αυτό μπορεί να γίνει πιο ελαφρύ με βάση την κατανομή της λίστας α, ε, της υπερεθνικής γιατί κατά την σύνθεση αυτής της λίστας, τα πανευρωπαϊκά κόμματα θα πρέπει να προσελκύσουν τους ψηφοφόρους τους. Τρία τέταρτα των πολιτών της Ένωσης ζουν στα 7 μεγαλύτερα κράτη-μέλη. Οι υπερεθνικές λίστες θα έχουν λοιπόν πολλούς υποψήφιους από τα μεγάλα κράτη-μέλη όπου ζουν οι ψηφοφόροι, ίσως όχι τα τρία τέταρτα, αλλά οπωσδήποτε όχι πολύ λιγότερο από το μισό. Κατ' ουσίαν, οι περισσότερες έδρες ε, θα καταληφθούν από υποψηφίους από τα μεγαλύτερα κράτη-μέλη. Και με αυτή την ανισορροπία αμφιβάλλουμε για το εάν οι ε, υπερεθνικές λίστες ε, θα αντέξουν πέρα από το 2019. Δεν μπορούν οπωσδήποτε να ανταγωνιστούν με την τέλεια λύση που προσφέρει η διπλή αναλογικότητα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πολύ. Ο καθηγητής συνοδεύεται και από τον κύριο Έλμπερμαν, ερευνητή από το Ίδρυμα Μαθηματικών του Augsburg. Μπορεί και αυτός να απαντήσει σε ερωτήσεις. Ας ακούσουμε τώρα τους ομιλητές και μετά να γίνει μια γενική συζήτηση για όλα τα θέματα. Περνάμε τώρα στον κύριο Μπρένταν Ολύρη που είναι καθηγητής πολιτικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο της Πενσιλβανίας αλλά επίσης και σύμβουλος της Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου και του ΟΗΕ. Ο καθηγητής Ολύρη έχει το λόγο. Χωρίς μικρόφωνο. Με μικρόφωνο. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ διαχωρίζω τις ε, συνομοσπονδιακές και ομοσπονδιακές προσεγγίσεις. Πρώτα την ομοσπονδιακή. Εδώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να ε, εφαρμόζει τις χωριστές ε, θέσεις των χωρών μελών γιατί δεν υπάρχει ενιαίος πανευρωπαϊκός λαός. Στην συνομοσπονδιακή προσέγγιση είναι ήδη υπερβολικά ομοσπονδιακό το κοινοβούλιο χωρίς να έχει την ανάλογη εντολή ή έγκριση από τις χώρες μέλη. Γιατί η συνταγματική συνθήκη απέτυχε. Επίσης δεν έχει δημοκρατική εντολή. Και αυτό φαίνεται και από την μεγάλη αποχή. Από το 79 που γίνονται άμεσες εκλογές συνεχώς πέφτει η συμμετοχή στις ευρωεκλογές και κάθε πέντε χρόνια οι φεντεραλιστές απογοητεύονται. Βέβαια αυξήθηκε λίγο η συμμετοχή γιατί αυξήθηκε ο πληθυσμός μετά την ένταξη των πρώην κομμουνιστικών χωρών αλλά υπάρχει εδώ ένα πανευρωπαϊκό φαινόμενο αποχής. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι 19 από τις 28 χώρες μέλη έχουν χαμηλότερη συμμετοχή στις εκλογές από τον μέσο όρο από τότε που εντάχθηκαν στην Ένωση. Αυτό βέβαια δεν λέει και πολλά για την ικανότητα κινητοποίησης του Spitzenkandidat. Όπως είπε μάλιστα ο καθηγητής Ματζόνη στην Ιταλία από το 2009 υπάρχει απόλυτο συσχετισμός μεταξύ δικαιοδοσιών του Κοινοβουλίου αυξανωμένων συνεχώς και μειωμένης συνεχώς συμμετοχής. Εγώ δεν νομίζω όμως ότι πρόκειται για αίτιο και αιτιατό, δηλαδή η μείωση των δικαιοδοσιών του Κοινοβουλίου δεν θα αύξανε τη συμμετοχή στις εκλογές. Παρόλα αυτά, ο συσχετισμό είναι ανησυχητικό και πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη από το Κοινοβούλιο. Αν πάρουμε στα σοβαρά την σπονδιακή συνταγή θα λέγαμε ότι δεν υπάρχει λόγο για ενιαίο εκλογικό νόμο, αλλά μάλιστα για την επαναφορά των ε, εκλογών στα εθνικά κοινοβούλια. Πέντε ωφέλη θα είχε αυτό. Πρώτον, κάθε μέλος του κοινοβουλίου θα είχε περισσότερη δημοκρατική νομιμότητα, διότι τα εθνικά κοινοβούλια ε, εκλέγονται με μεγαλύτερη συμμετοχή. Έπειτα, οι ευρωβουλευτές θα έχουν την ίδια εντολή με τα εθνικά κοινοβούλια και δεν θα υπάρχουν επομένως επικαλύψεις και αντιφάσεις πράγμα που συμβαίνει συχνά γιατί είναι διαφορετική η εκλογική κύκλη των ευρωεκλογών και των εθνικών κοινοβουλίων. Τρίτον, οι Ευρωπαίοι πολίτες θα έχουν μία λιγότερη εκλογή κάθε πέντε χρόνια και αυτό θα αύξανε τη συμμετοχή. Τέταρτον, αυτή η μετάβαση, η επιστροφή στον κόσμο πριν το 79 μπορεί να οθούσε την δημοκρατική νομιμότητα των Ευρωβουλευτών με μεγαλύτερη σύνδεση μεταξύ εθνικών κομμάτων και βουλών γιατί θα υποχρεωνόταν τα, οι βουλές να οργανώνονται πολύ καλύτερα να οργανώνουν πολύ καλύτερα τα ευρωπαϊκά θέματα τους και έτσι θα μειωνόταν το δημοκρατικό έλλειμμα με την αύξηση των δικαιοδοσιών των εθνικών βουλών. Βέβαια, κάθε τέτοια αντιδραστική, όπως θα λέγαμε, αντιμετώπιση θα είχε και δυσκολίες. Ιδιαίτερα το ότι δεν χρησιμοποιούν όλα τα κράτη την αναλογική στις εκλογές, εκτός από, στις ευρωεκλογές, εκτός από τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Θα μπορούσαν όμως να οθηθούν να το πράξουν, ίσως χωριστό ψηφοδέλτιο για τους ευρωβουλευτές ή κυρώσεις αν δεν χρησιμοποιείται η αναλογική στις ευρωεκλογές. Βέβαια μια τέτοια αλλαγή θα σήμαινε και ότι οι ευρωβουλευτές μπορεί να έχουν επικαλυπτόμενα καθήκοντα εθνικά και ευρωπαϊκά και με μεγαλύτερο κόστος για την ενοικίαση σπιτιών κλπ. Αλλά θα μπορούσε να υπάρξει καλύτερο συντονισμός και τουλάχιστον να καταργηθεί το Κοινοβούλιο του Στρασβούργου που δεν έχει καμία δικαιολόγηση εκτός από το ότι το λένε οι συνθήκες. Τρίτον, οι εντολές, αν γινόταν αυτή η επιστροφή των εκλογών στα εθνικά κοινοβούλια, θα απλοποιούσαν πολλά πράγματα. Υπάρχει αυτό και σε άλλα συστήματα. Μπορεί να λυθεί το πρόβλημα με την σύγκληση του ρυθμού των εκλογών πανενωσιακός ας πούμε τετραετή εκλογικό κύκλο Άλλη δυσκολία θα ήταν εάν οι χώρες μέλη θα συνέχιζαν ή όχι να εφαρμόσουν διαφορετικές μορφές αναλογικής εκπροσώπησης. Ήδη αυτό συμβαίνει στα Εθνικά Κοινοβούλια, δεν είναι δηλαδή ιδιαίτερο πρόβλημα και για, το συνομοσπονδιακό, για τη συνομοσπονδιακή προσέγγιση. Καλό θα ήταν νομίζω να σκεφτούμε στη Θεσμική Επιτροπή ότι υπάρχει σοβαρό θέμα εξέτασης της συνομοσπονδιακής προσέγγισης. Δεν είναι τίποτε τρελό και παράλογο και θα μπορούσε να προωθηθεί από όσους είναι υπέρ της Ένωσης, όχι μόνο από τους ανθενωτικούς. Θα μπορούσαμε να το δοκιμάσουμε αυτό σε δημοψηφίσματα την ιδέα για να δούμε αν οι πολίτες προτιμούν άμεσες ή έμεσες ευρωεκλογές να δοκιμάσουμε αν το κοινό είναι υπέρ της εθνικής ευρωεκλογής ή της υπερεθνικής. Θα μπορούσε να δοκιμαστεί το σύστημα της εκλογής διακλήρου. Αλλά καταλαβαίνω ότι οι περισσότεροι από εσά και οι περισσότεροι ευρωβουλευτές είναι μάλλον φεντεραλιστές και όχι Συνομοσπονδιακοί Θεωρούν ότι πρόκειται εδώ για το κοινοβούλιο μιας ομοσπονδίας και άρα πρέπει να εκλέγεται χωριστά. Υπάρχουν όμως ομοσπονδίες που δεν έχουν ενιαία εκλογική διαδικασία. Μπορούν να λειτουργήσουν και χωρίς αυτήν. Είναι φανερό ότι η ενιαία εκλογική διαδικασία θα καθιστούσε πιο φεντεραλιστική την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά ποιο θα ήταν το αποτέλεσμα ως προς τη δημοκρατική νομιμότητα και ιδιαίτερα ως προς τη μείωση της αποχής στις ευρωεκλογέ. Τρεις παράγοντες επηρεάζουν τη συμμετοχή στις εκλογές. Ένα, μπορεί να αυξηθεί η συμμετοχή με την υποχρεωτική ψηφοφορία, αλλά το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή σας δεν έχουν τη δημοκρατική νομιμότητα, ίσως όχι και τη δικαιοδοσία να επιβάλλουν υποχρεωτική ψηφοφορία. Δεν είναι τίποτε αντιδημοκρατικό βέβαια η υποχρεωτική ψηφοφορία, αλλά δυστυχώς πολλές από τις πρώην κομμουνιστικές χώρες δεν θα το δέχονταν και 87% παραδείγματος χάρη των Σλοβάκων ενθουσιαστικά θα ήθελαν να μην είναι υποχρεωτική η ψηφοφορία. Πάντως είναι συμβατή με τη, δημοκρατία. Φαντάζομαι όμως ότι δεν το σκέφτεστε καν. Οι δύο άλλοι παράγοντες που θα μπορούσε να εφαρμόσει το Κοινοβούλιο για να αυξηθεί η συμμετοχή είναι πρώτον η διασφάλιση του ότι οι εκλογές θα γίνονται την ίδια μέρα με τις εθνικές. Βέβαια δεν αρέσει αυτό σε όλους τους φεντεραλιστάς, διότι θέλουν χωριστή εντολή για το Ευρωκοινοβούλιο, αλλά θα μπορούσε αυτό να αυξήσει τη συμμετοχή μεταξύ 10 και 20% παραπάνω για τις χώρες που δεν έχουν υποχρεωτική ψηφοφορία. Και ο τρίτος παράγοντας που θα μπορούσε να αυξήσει τη συμμετοχή είναι μαζική επέκταση των δικαιοδοσιών της Ένωσης και του Κοινοβουλίου για θέματα κράτους ευημερίας, θεμάτων πολέμου και ειρήνης κτλ. Φυσικά αυτό θα αύξανε τη συμμετοχή, αλλά φυσικά δεν υπάρχει εντολή για κάτι τέτοιο. Επομένως αυτό που συστήνω είναι ότι υπάρχουν πολύ λίγοι τρόποι, ίσως και κανείς, για να μπορέσει το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή σας να αυξήσει σημαντικά τη συμμετοχή στις ευρωεκλογέ. Εν μέρη διότι όλα τα κράτη-μέλη τώρα έχουν εγκρίνει την αναλογική εκπροσώπηση και οποιοδήποτε μεγαλύτερο κίνητρο για συμμετοχή δεν υπάρχει πια. Το θέμα αντίθετα είναι ποια αναλογική εκπροσώπηση είναι η καλύτερη. Και εδώ νομίζω ότι είναι σαφές, μπορώ να σας πω με βεβαιότητα, ότι υπάρχει συνένεση μεταξύ των πολιτικών επιστημόνων ως προς το ποια αναλογική, ποιο αναλογικό σύστημα είναι το καλύτερο. Για την αύξηση της συμμετοχής, τα κίνητρα που δίνονται στους εκλογείς, όπως το ενιαίο σύστημα μεταφοράς ψήφου, θα ήταν σοβαρό επιχείρημα για τα ανοιχτά ψηφοδέλτια και θα μπορούσε να αυξήσει λιγάκι τη συμμετοχή από ότι τα κλειστά. Η μεικτή αναλογικότητα όπως χρησιμοποιεί η Γερμανία θα ήταν η δεύτερη ή τέταρτη επιλογή, δεύτερη, τρίτη ή τέταρτη επιλογή. Από την άποψη της πολιτικής επιστήμης είναι ότι τα εκλογικά συστήματα τελικά όποια και να είναι δεν έχουν πολύ διαφορετικά αποτελέσματα το ανοιχτό με το κλειστό πληφοδέλτιο δεν έχουν τρομερή διαφορά στο αποτέλεσμα νομίζω ότι θα ήταν λάθος είτε είναι κανείς συνομοσπονδιακός είτε ομοσπονδιακός να οθήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση σε μία ενιαία μορφή αναλογικής εκπροσώπησης και θα ήταν ιδιαίτερα λάθος η Ιρλανδία και η Μάλτα, η Ιρλανδία και Βορράς και Νότος που χρησιμοποιούν το σύστημα που χρησιμοποιούν να υποχρεωθεί να μεταφέρει τους υποψηφίους της σε άλλες χώρες. Θα θεωρούνταν απαράδεκτο. Μια άλλη μέθοδος θα ήταν η αύξηση της δραστηριότητας ευρωπαϊκών κομμάτων. Μελικοί θέλουν να μειωθεί ο κατακαιρματισμός έτσι μεταξύ του Κοινοβουλίου μέσω της δημιουργίας υπερεθνικών κομμάτων ή αν μεγαλύτερου ορίου για τη συμμετοχή των κομμάτων. Αν επιβληθούν τέτοια όρια, μπορεί περιφερειακά να αλλάξει η συμμετοχή, αλλά περιφερειακά. Γιατί είναι γνωστό ότι δεν αυξάνεται δραματικά η συμμετοχή με αυτό το κριτήριο. Εξάλλου είναι φανερό ότι η ψηφοφορία τα Σαββατοκύριακα ευνοεί τη μεγαλύτερη συμμετοχή, αλλά μάλλον δεν πρόκειται να καθοριστεί μία ενιαία ημέρα για ψηφοφορία για όλη την Ένωση, ούτε θα έχει σημαντικά αποτελέσματα ως προς την αποχή. Θα ήταν μάλλον συμβολικό μέτρο. Συμφωνώ ότι πρέπει να ερευνηθούν περισσότερο όλα αυτά και να, η δυνατότητα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, ιδιαίτερα για το κατά πόσον είναι ασφαλής ή όχι. Και αυτό με δημοψηφίσματα για να δούμε τι ηλεκτρονικά ψηφοδέλτια θα μπορούσαν να δουλέψουν καλύτερα. Άλλο θέμα που πάντοτε αντιμετωπίζει το Κοινοβούλιο είναι με τι να συγκριθεί. Και το πρωί πρώτη ομιλία έλεγε ότι πρέπει να μην ανησυχούμε για τη χαμηλή συμμετοχή στι ευρωεκλογέ, διότι το ίδιο συμβαίνει και με τις τοπικές και περιφερειακές εκλογές ολόκληρη την Ευρώπη. Γενικά όμως το Κοινοβούλιο θεωρεί τον εαυτό του ως φεντεραλιστικό όργανο και συγκρίνεται με τα εθνικά. Αν συγκρίνουμε τη συμμετοχή στις, εκλογές, με τις εθνικές και με ομοσπονδιακές δημοκρατίες παγκοσμίω, είναι φανερό ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει από τις μεγαλύτερες αποχές και μπορεί να συγκριθεί μόνο με την Ελβετία και τις Ηνωμένε Πολιτείες. Όταν στις Ηνωμένε Πολιτείες ε, η Βουλή των Αντιπροσώπων εκλέγεται σε περίοδο τουλάχιστον που δεν ταυτίζεται με την εκλογή της προεδρικές. Και το κοινό που έχει ένωση με την Ελβετία και τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι η πολυπλοκότητα του φεντεραλιστικού συστήματος, πολλές εκλογές και δεν υπάρχουν δεν είναι καθοριστικός ο, η καθοριστική ψήφος των πολιτών για την τύχη της Ομοσπονδίας. Αυτά όλα εξηγούν την μεγάλη αποχή παραπάνω από άλλους παράγοντες που θα μπορούσε κανείς να φανταστεί. Επειδή λοιπόν το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή σας κυριαρχείται από εκείνους που έχουν φεντεραλιστικές απόψεις αυτό που θα έπρεπε να αποφευχθεί στο μέλλον είναι το εξής να μην ζητηθεί ενιαία αναλογική εκπροσώπηση. Δεν υπάρχει συνένεση επιστημονική επ' αυτού. Υπάρχει πολύ μεγαλύτερη συνένεση για τα υπάρχοντα συστήματα όπου κυριαρχεί όποιος έχει πάρει τους περισσότερους ψήφους και πρημοδοτείται. Δεύτερον, νομίζω ότι δεν πρέπει να υπάρχει ενιαίος εκλογικός νόμος, αλλά μάλλον να προσπαθήσει το Κοινοβούλιο να προωθήσει βέλτιστες πρακτικές <coughs> στην Ένωση μεταξύ των οποίων και καλύτερη εκπροσώπηση των γυναικών, εθνικών μειονοτήτων και μεταναστών. Τρίτον, θα ήταν νομίζω λογικό για το Κοινοβούλιο να αποφύγει διαμάχες με εθνική νομοθεσία για την ηθαγένεια. Ταυτόχρονα όμως να προωθήσει βέλτιστες πρακτικές. Παραδείγματος χάρη να έχουν το δικαίωμα και οι ξένοι σε μια χώρα να ψηφίζουν στις ευρωεκλογέ τουλάχιστον. Αυτό δεν επιτρέπεται από όλες τις χώρες. Είναι και αυτό μια σύσταση βελτίστων πρακτικών. Πολύ πιο, με πολύ λιγότερη συνένεση είναι, θα ήταν οι επιπτώσεις εκλογών για το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Τα δικαστήρια πολλές φορές ε, κάνουν συμβιβασμούς για πολιτικούς λόγους. Ας πούμε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων θεώρησε απαράδεκτη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση ε, τη συλλογική προεδρία στη Βοσνία Ερζεγοβίνη και τη διαδικασία εκλογών της Γερουσίας εκεί. Ό,τι και να πούμε για την απόφαση αυτή, το δικαστήριο κατήργησε ένα συνταγματικό εκεί δικαίωμα και ζήτησε να μην γίνεται σεβαστό ένα δικαίωμα εκεί. Σήμερα στην Επιτροπή σας ένα από τα προβλήματα είναι ότι το Γερμανικό Συνταγματικό Δικαστήριο έχει συγκεκριμένη άποψη για τα εκλογικά όρια με τα οποία διαφωνούν πολλοί ευρωβουλευτές και πολλές χώρες. Σκεφτείτε το καλά. Θέλετε να δώσετε δικαιοδοσίε στα δικαστήρια, αν το κάνετε αυτό θα υπάρξουν ίσως αρνητικές και μακροχρόνιες συνέπειες γιατί τα δικαστήρια πάντοτε αποφασίζουν με τρόπο που πρέπει να γίνεται σεβαστή η απόφαση τους, ό,τι και να είναι. Είναι λοιπόν λογικό να υπάρχει με, με ένας διαφανής κανόνας για την ε, εκπροσώπηση, αλλά χάρη της διαφανίας θα ήταν πολύ καλύτερο να εκφραστούν όλα αυτά μέσω ορισμένων απλών αρχών ελαχίστων ορίων εκπροσώπησης από τις χώρες μέλη και όχι των υψηλότερων ορίων όπως οι κανόνες δοχών για την αναλογική εκπροσώπηση. Ενδιαφέρον είναι να δούμε τη σύνδεση μεταξύ εκλογικών διευθετήσεων για το Κοινοβούλιο και δικαιοδοσιών των κρατών μελών στο Συμβούλιο. Αν η Ένωση θέλει ποτέ να λειτουργήσει ως Ομοσπονδία, τότε το λογικό θα ήταν να κινηθεί προς αναλογικότητα στο Κοινοβούλιο με ισότητα μεταξύ των χωρών μελών στο Συμβούλιο. Αν δεν γίνει κάτι τέτοιο θα, είναι, θα πρόκειται πάντοτε για ένα ατυχή συμβιβασμό δύο ειδών αναλογικότητας με δύο μέτρα και δύο σταθμά. Στα δύο αυτά όργανα της Ένωσης. Από τη θετική μεριά θα έλεγα ότι η Θεσμική Επιτροπή μπορεί να πρέπει να εξετάσει το κατά πόσον οι ευρωβουλευτές θα έπρεπε να εκλέγονται μεταξύ των εθνικών βουλευτών ή από ανεξάρτητους υποψήφιους. Αυτό που λέμε σορτήσιον εμείς. Εγώ δεν πιστεύω ότι οι προτάσεις για υπερεθνικά ψηφοδέλτια ή για δεύτερο επίπεδο προσώπηση είναι σωστές. Δεν είναι σωστές διότι πρώτον καταπολεμούν τη λογική της αναλογικής εκπροσώπησης που σημαίνει ακριβώς ότι τα κράτη-μέλη θα έχουν την εγγύηση ότι θα έχουν έναν προβλέψιμο αριθμό ευρωβουλευτών. Η τα υπερεθνικά ψηφοδέλτια ε, κάνουν όλα αυτά τα πράγματα απρόβλεπτα και άρα υπονομεύουν το ίδιο το εκλογικό συμβόλαιο με τους πολίτες. Έπειτα νομίζω ότι οι πολιτικές ταυτότητες δεν υπάρχουν για να δημιουργηθούν όντως υπερεθνικά ψηφοδέλτια και πρέπει να αποφύγουμε τους τεχνητούς μηχανισμούς που θα μπερδέψουν το κοινό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ καθηγητή Ολύρη. Νομίζω ότι θα γίνει Πολύ συζήτηση να, με βάση την παρουσίασή σας να ζητήσω από τον καθηγητή Ρομπέρτο Νταλιμόντε που είναι από το ε, Πανεπιστήμιο της Φλωρεντίας αλλά διδάσκει και στη Νέα Υόρκη. Παρακαλώ. I'm going to show some data. Θα σας δείξω κάποια στοιχεία. Oh. I hope they are visible. Ελπίζω να φαίνονται. Since the, uh, it's, it's, uh, it's a big, yes, that's the reason I said I hope they are visible. Ελπίζω λοιπόν να φαίνεται γιατί είναι μικρά εδώ στη διαφάνεια. Είναι με μικρούς χαρακτήρες. Εδώ έχουμε τα 28 εκλογικά συστήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και σαφώς η εικόνα δεν παρουσιάζει ομοιομορφία. Το πρώτο ερώτημα λοιπόν Δεν δουλεύει και το λέιζερ. Α, όχι, δουλεύει. Δεν είναι μία εικόνα λοιπόν, σε καμία περίπτωση. Και το πρώτο ερώτημα που τίθεται είναι πώς μπορούμε να επιτύχουμε ομοιομορφία. Εγώ θα έλεγα ότι η ομοιομορφία, εάν είναι επιθυμητό, θα μπορούσε να ε, επιτευχθεί στη στήλη που έχουμε την ε, ε, ηλικία. Πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να ενερμονίσουμε τουλάχιστον κάποια πράγματα, αλλά εκεί που μας ενδιαφέρει περισσότερο είναι τι έχουμε στις άλλες στήλε. Εδώ έχουμε ε, την αναλογική εκδοχή που χρησιμοποιεί το κάθε κράτος μέλος. Εγώ προσωπικά δεν νομίζω ότι θα αλλάξει και τίποτα αν έχουμε ομοιομορφία ή όχι. <laughs> Οι διαφορές προκύπτουν από την αναλογικότητα ή την έλλειψη αναλογικότητας του συστήματος. Επομένως δεν έχει καμία σημασία. Η την ελλειψη αναλογικοτητας του συστηματος οποτε δεν αυτή που αναφέρει τις μεθόδους επιλογής ε, υποψηφίων έχω βάλει εδώ στήλο ε, preferential voting, αλλά στην πραγματικότητα είναι σύστημα. Έχουμε λίστες και ψηφοδέλτια. Πρόκειται για ανοιχτά ψηφοδέλτια, αλλά διαφορετικά, διαφορετικές μορφές ανοιχτών ψηφοδελτίων. Και εδώ είναι ένα σημείο στο οποίο θα μπορούσαμε να έχουμε μία συζήτηση για το κατά πόσον η ομοιομορφία ή τουλάχιστον η μεγαλύτερη εναρμόνιση θα αυξήσει και τη νομιμοποίηση ή τη συμμετοχή στις ευρωεκλογές. μέσω καλύτερης προσέγγισης των υποψηφίων. Ε, θα δείτε ότι από τις λίγες χώρες που έχουν ε, ε, λίστα, ε, έχουμε πολύ μικρές, μικρό αριθμό χωρών, οι περισσότερες έχουν ανοιχτά ψηφοδέλτια. Κυρίως μας ενδιαφέρει όμως η προηγούμενη στήλη, η στήλη που έχει τα κατώτατα όρια και είναι και ε, η στήλη που έχει και το μέγεθος των εκλογικών περιφερειών. περιφερειών. Εννέα χώρες, είναι πιο εύκολο ίσως να τα δούμε με αυτή τη διαφάνεια, εννέα χώρες δεν έχουν καθόλου ε, κατώτατο όριο για να εκλεγεί κάποιος και εδώ έχουμε χώρες που έχουν 5% ε, όριο στην αριστερή στήλη και κάποιες που έχουν λίγο μικρότερο στη μέση. Εδώ βέβαια είναι και ένας τομέας όπου θα μπορούσαμε ίσως να έχουμε μεγαλύτερη εναρμόνιση ή ομοιομορφία. Ακόμα και έτσι, και πάλι δεν θα καταφέρουμε να έχουμε ένα ομοιόμορφο εκλογικό σύστημα, διότι η πλήρης ομοιομορφία δεν μπορεί να επιτευχθεί εδώ ε, λόγω των περιφερειών, λόγω του μεγέθους των διαφόρων περιφερειών, διότι όπως γνωρίζετε αυτό σχετίζεται με τον αριθμό των εδρών που ε, λαμβάνει κάθε χώρα μέλος. Και αυτό φυσικά δεν μπορεί να εναρμονιστεί. Because of Λόγω αυτών των περιορισμών, το αποτέλεσμα που θα έχουμε θα είναι μάλλον κάτι που ομοιάζει με αυτή τη διαφάνεια. Εδώ έχω βάλει σε μια κλίμακα 7 ε, βαθμών ε, αυτή την έλλειψη αναλογικότητας των 28 εκλογικών συστημάτων. Πάμε από πολύ χαμηλή, δηλαδή αυτά είναι τα πιο αναλογικά συστήματα, το σύστημα της Γερμανίας και της Ισπανίας, Έχουμε λοιπόν το σύστημα το οποίο είναι υψηλά αναλογικό και φτάνουμε σε ένα τελείως ε, δυσανάλογο, χωρίς καμία αναλογική ψήφο, την Ιρλανδία και την Πολωνία και όλες οι υπόλοιπε χώρες είναι στη μέση. Αν αλλάξουμε λίγο τα κατώτερα τα όρια, θα μπορούσαμε ίσως να αλλάξουμε λίγο την κατάσταση σε κάποιο βαθμό, αλλά όχι οριστικά, διότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα για το ε, μέγεθος της εκλογικής περιφέρειας. Ακόμα και αν θεωρήσουμε ότι θα μπορούσαμε να μειώσουμε τα κατώτατα όρια εισαγωγή ε, ή να τα διαγράψουμε εντελώ και πάλι θα έχουμε αποτελέσματα χωρίς αναλογικότητα στα περισσότερα κράτη-μέλη λόγω του διαφορετικού μεγέθους των εκλογικών περιφερειών. Κατόπιν τούτου, θα ήθελα να θέσω το εξής ανησυχητικό ερώτημα. Χρειαζόμαστε πραγματικά ομοιομορφία. Γιατί αναφερόμαστε σε έναν ενιαίο εκλογικό νόμο. Τι σκοπό εξυπηρετεί ένας ενιαίος νόμος. Εγώ δεν έχω καταλάβει και νομίζω ότι θα πρέπει να το διευκρινίσουμε. Διότι εάν ο σκοπός μιας ενιαίας εκλογικής διαδικασίας είναι να αυξηθεί η νομιμοποίηση και η συμμετοχή στις εκλογές και τα δύο ε, σε κάποιες περιπτώσεις, νομίζω ότι απατώμεθα όλοι ικτρά. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να αυξηθεί η συμμετοχή και μάλιστα δεν θα αυξηθεί και καθόλου με ενιαία εκλογική διαδικασία. Αν πραγματικά πιστεύουμε ότι χρειαζόμαστε έναν νέο εκλογικό νόμο, για οποιοδήποτε λόγο που δεν ε, μπορώ να αντιληφθώ ποιος είναι αυτή τη στιγμή, νομίζω ότι η πρόταση Μπούκεσχάιμ είναι, ε, είναι ενδιαφέρουσα. Να πω όμως κάτι που γνωρίζω ότι ξέρουν ε, ο καθηγητής Πόκελσχάιμ και η ε, κυρία Όμπερ Μάιερ. Εάν περάσουμε από ένα εκλογικό σύστημα σαν αυτό που έχουμε και περάσουμε στην πρόταση Πόλκενσχάιμ, προκύπτει το εξή. Η διπλή αναλογικότητα πληρεί δύο προϋποθέσεις. Την προϋπόθεση ότι τα κράτη-μέλη θα λάβουν τις έδρες που τους αναλογούν και ότι τα κόμματα θα λάβουν τις έδρες που τους αναλογούν σε αναλογική βάση, αλλά υπάρχει και μια τρίτη συνιστόσα που δεν είναι μαθηματική προϋπόθεση και πρέπει ε, να πληρείται βάση του συστήματος. Είναι μια πολιτική προϋπόθεση. Και αυτό είναι το γεγονό ότι τα κόμματα εκλέγουν ε, υποψηφίους όταν λάβουν τις περισσότερες ψήφους. Και εδώ υπάρχει ένα τεχνικό ζήτημα. Στην Ιταλία προσπαθούμε να κάνουμε μεταρρύθμιση του εκλογικού νόμου και αντιμετωπίσαμε το συγκεκριμένο πρόβλημα, διότι αυτό συμβαίνει με αυτά τα συστήματα. Οι υποψήφοι μπορούν να εκλεγούν, υπάρχουν προϋποθέσεις, μέσα στην ίδια λίστα ε, όπου μπορεί να εκλεγεί κάποιος με λιγότερες ψήφους σε σχέση με έναν υποψήφιο που βρίσκεται σε άλλη λίστα, σε άλλη περιφέρεια. Mm-hmm. Και αυτό λοιπόν είναι ένα πιο πολιτικό ζήτημα, δεν είναι περισσότερο μαθηματικό. Από πολιτική σημασία όμως έχει μεγάλη ε, βαρύτητα. Ναι. Η πρόταση Πόλκενσχάιμ, οι αντίστοιχε προτάσει ε, για τη δημιουργία εκλογικών συστημάτων που θα είναι αποτελεσματικά σε επίπεδο ένωση, ε, προϋποθέτουν την ύπαρξη υπερεθνικών κομμάτων που ε, ανταγωνίζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και όχι σε εθνικό επίπεδο. Μόλις ακούσαμε τις επικρίσεις από τον καθηγητή Ολύρη για τη δημιουργία και την προώθηση ε, αυτών των υπερεθνικών κομμάτων και της λίστας της αντίστοιχης. Ανεξάρτητα όμως από αυτές τις επικρίσεις που μόλις άκουσα, θα ήθελα να πω κι εγώ κάτι από αυτού, που ξέρω ότι είναι ευσεβής πόθος μεν, αλλά καλό είναι καμιά φορά να σκεφτόμαστε και λίγο πιο μακρόπνοα. Να σας πω καταρχάς ότι τα συστήματα αναλογικής εκπροσώπησης, που είναι τα συστήματα που έχουμε τη σήμερα ημέρα, δεν περιλαμβάνουν κανένα κίνητρο για τη δημιουργία υπερεθνικών ε, ψηφοδελτίων. Στα υπερεθνικά ψηφοδέλτια θα υπάρξουν μόνο εάν υπάρξουν κάπου κίνητρα. Επομένως, συστήματα ομοίων, ε, σαν αυτά που έχουμε εμείς, δεν παρέχουν κανένα κίνητρο. Το όριο που προτείνει ο καθηγητής Πολκενσχάιμ ε, είναι ένα, ένα σχετικό κίνητρο. Ένα άλλο κίνητρο θα μπορούσε να είναι η δημόσια χρηματοδότηση ε, αυτών των υπερεθνικών κομμάτων και των αντίστοιχων ψηφοδελτίων και ένα άλλο ενδιαφέρον κίνητρο θα μπορούσε να προκύψει εάν ε, προχωρήσουμε την πρόταση DAF. Η πρόταση DAF, που, όπως μόλις ακούσαμε, προϋποθέτει τη δημιουργία 25 ευρώ που θα δίνονται σε ε, επίπεδο ένωσης σε μια ευρωπαϊκή εκλογική περιφέρεια ένα ψηφοδέλτιο επικρατεία ουσιαστικά. Υποθέτω ότι αυτές οι θέσεις θα δίνονται αναλογικά. Τι γίνεται αν δίνονται ως μπόνους για το υπερεθνικό ε, ε, ψηφοδέλτιο, για το Ευρωπαϊκό Κόμμα ή για ένα συνασπισμό ευρωπαϊκών κομμάτων που θα αποκτήσουν την πλειοψηφία των ψήφων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σας είπα απλώ ότι αυτό είναι ευσεβής πόθος, έτσι. Λόγω της κατάστασης των ευρωπαϊκών υποθέσεων. Ήθελα όμως να τη θέσω αυτή την πρόταση, διότι μέσω της δημιουργίας αυτών των ε, εδρών ε, ε, μπόνους που θα πάει ναι, στα κόμματα που θα πάρουν τις περισσότερες ψήφους σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ουσιαστικά παρέχουμε πολύ ισχυρά κίνητρα για τη δημιουργία αυτού του υπερεθνικού ψηφοδελτίου. Αλλά υπάρχει και το εξή ε, σε αυτή την πρόταση. Κατά την άποψή μου, ο πραγματικός λόγος για τον οποίο είναι μικρή συμμετοχή στις εκλογές είναι γιατί οι Ευρωπαίοι ψηφοφόροι θεωρούν ότι αυτές οι εκλογές δεν έχουν καμία σημασία και θεωρούν ότι δεν έχουν καμία σημασία διότι οι εξουσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι είτε ισχυρέ είτε πολύ αδύναμε. Δεν έχουν σημασία γιατί οι Ευρωπαίοι ψηφοφόροι δεν θεωρούν ότι αυτέ οι εκλογέ είναι αποφασιστική σημασία. Δεν θεωρούν ότι διακυβεύεται κάτι. Τι διακυβεύεται σε κάθε ε, τέτοια εκλογική αναμέτρηση. Το να είναι λοιπόν πιο σημαντικές οι ευρωεκλογές είναι το κλειδί για να έχουμε ίσως αύξηση της συμμετοχής. η αποφασιστική σημασία των εκλογών είναι μια πολυδιάστατη έννοια, την οποία δεν έχω το χρόνο εδώ να ε, σας αναπτύξω διεξοδικά, αλλά εάν ε, προχωρήσουμε λίγο την πρόταση DAF και έχουμε αυτές τις έδρες ως μπόνους, ίσως θα είναι μια ιδέα, θα δημιουργήσει την εντύπωση στους ψηφοφόρους ότι διακυβεύεται κάτι και ότι ε, θα ενισχυθεί αυτό μέσω των ε, καλύτερων των κομμάτων σε αυτή τη λίστα για αυτές τις έδρες. Ε, όπως είπατε και εσείς κύριε Ντάφ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ καθηγητή Ταλιμόντε. Να δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Μπερτοντσίνη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Παίρνω το λόγο τελευταίος. Γεγονός το οποίο μου επέτρεψε να ακούσω και να συμφωνήσω με πολλά από αυτά τα οποία ακούστηκαν και θα ε, ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να προσθέσω κάτι για να διευρύνουμε τη συζήτηση. Ξεκινώ από ένα λίγο διαφορετικό πρίσμα. Ε, γιατί να πρέπει να μεταρρυθμίσουμε την εκλογική διαδικασία. Ε, όταν ήρθα εδώ, ε, απαντώντας την ευγενική σας πρόσκληση, Είπα εντάξει να έρθω, αλλά για ποιο λόγο θέλουμε να μεταρρυθμίσουμε την εκλογικό νόμο. Θα σταθώ λίγο στους στόχους λοιπόν και από εκεί και πέρα θα δω τι μπορούμε να κάνουμε όσον αφορά τις βασικές προτεραιότητες. Νομίζω ότι αυτό γίνεται σε ένα πολιτικό πλαίσιο το οποίο ε, περιέχει μια καινοτομία. Αυτή τη διαδικασία του Spitzenkandidat, ε, του επικεφαλής του ψηφοδελτίου υποψηφίου για την ε, Προεδρία τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κάτι το οποίο ήταν πολύ θετικό για μας και μας επέτρεψε να δώσουμε ένα πρόσωπο στην πολιτική δομή της λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά και του πολιτικού βίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και θεωρώ ότι από εκεί θα πρέπει να ξεκινήσουμε. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο εκπροσωπεί τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, θέλει να δώσει πρόσωπο, να ε, ε, υπάρχει ένα, μια φυσιογνωμία που να ανταποκρίνεται σε αυτό το οποίο θεωρούν ως ευρωπαϊκό. Αυτό το οποίο μας επέτρεψε αυτή η διαδικασία του Spitz candidat να βελτιώσουμε είναι ότι επιτρέπει να δούμε σε τι θεμελιώνονται οι ελπίδες των Ευρωπαίων πολιτών και ε, τι πρεσβεύουν, με ποια ιδεολογία συμφωνούν. Καταρχάς, θεωρώ ότι αυτό θα πρέπει να είναι ο βασικός στόχος λοιπόν της μεταρρύθμισης τη εκλογική διαδικασία. Υπάρχουν και δευτερεύοντες ε, στόχοι, τους οποίους θα προσπαθήσω να σας αναπτύξω αργότερα. Θεωρώ ότι ίσως θα έπρεπε να προσαρμόσουμε και τη διαδικασία βάσει αυτών. Καταρχάς, όμως, οι στόχοι της μεταρρύθμισης κατά την άποψή μου, δεν μπορούν να είναι ένας πρώτος στόχος που για μένα είναι δευτερεύον, η αύξηση της συμμετοχή της ευρωεκλογέ. Δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι αυτός ο στόχος, διότι η συμμετοχή καταρχάς δεν σχετίζεται με θεσμικά στοιχεία. Η συμμετοχή σχετίζεται με συνταγματικά στοιχεία. Νομίζω ότι το είπε προηγουμένως και ο κύριος Ολύρη υπάρχει ένα έλλειμμα αρμοδιοτήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνολικό έλλειμμα. Είμαστε σε ε, πεδίο επικουρικότητας. Επομένως, το ποσοστό της συμμετοχής σχετίζεται με αυτό το έλλειμμα, το σχετικό έλλειμμα αρμοδιοτήτων. Εάν οι αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυξηθούν σημαντικά, τότε μπορεί να αυξηθεί και η συμμετοχή. Αλλά ε, αν αναφερόμαστε στο ποσοστό τη συμμετοχή στι ευρωεκλογέ, όπως είπε ο κ. Σολίδη, και το ε, ποσοστό των, ε, ε της συμμετοχής στη, στην Ελβετία ή στην Αμερική, στι ομοσπονδιακέ εκλογές, τότε θα δούμε ότι λίγο πολύ στα ίδια είμαστε ε, υπάρχει αυτός ο μύθος ότι, ότι ε, το 80% της εθνικής νομοθεσίας προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι όμως το 80% της εθνικής νομοθεσίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γι' αυτό και ακριβώς είναι μικρή συμμετοχή. Αν θέλουμε να είμαστε πιο αντικειμενικοί, υπάρχει μια καλή συμμετοχή, η οποία θα μπορούσε να βελτιωθεί και θα βελτιωθεί την ημέρα όχι ε, οι εξουσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα αυξηθούν, αλλά οι αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα είναι αυτές που θα αυξηθούν. Αλλά για να αυξηθούν δεν μπορούμε να λέμε ότι το 80% της νομοθεσίας που έχουμε σε εθνικό επίπεδο προέρχεται από τις Βρυξέλλες γιατί δεν θα ήταν σωστό. Τώρα, το γεγονός ότι ο κόσμος πηγαίνει να ψηφίσει είναι ότι υπάρχει συγκεκριμένο πλαίσιο. Σε αυτές τις εκλογές είχαμε κρίση την εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το γεγονός ότι θα μπορούσαν να έχουμε και τοπικές και εθνικές εκλογές την ίδια ημέρα. Αυτό μπορεί να συνεισφέρει. Θα μπορούσαμε να κάνουμε και περισσότερο, να δώσουμε δικαίωμα ψήφου στους Ευρωπαίους και στη χώρα καταγωγής και όχι στη χώρα ε, στην οποία ζουν, να υπάρχει ε, και ηλεκτρονική δυνατότητα ψήφου. Ε, αλλά δεν θα πω άλλα τώρα εδώ. Νομίζω ότι ε, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η κατάσταση είναι ίσως απελπιστική, αλλά όχι πάρα πολύ σοβαρή. Δεν θα πρέπει όμως η αύξηση της συμμετοχής να είναι στόχος της μεταρρύθμισης της εκλογικής νομοθεσίας. Δεύτερος στόχος που είναι πιο χρήσιμος από τον πρώτο, αλλά και πάλι είναι δευτερεύον, είναι να διορθώσουμε το θέμα της κατανομής των εδρών μεταξύ των κρατών μελών. Εγώ είμαι υπέρ φυσικά της διόρθωσης. Αν μπορέσουμε να ε, υιοθετήσουμε και το μοντέλο CAMCOM, ίσως θα ήταν πιο δίκαια ε, τα πράγματα και θα χρειαζόντουσαν και κάποιες ε, ε, μικρές διορθώσεις, αλλά θα ήταν καλύτερη από την κατάσταση που έχουμε αυτή τη στιγμή. Η κατάσταση είναι ότι δεν έχουμε δυνατότητα να ε, αλλάξουν τα πράγματα λόγω της ψήφου ενός ψηφοφόρου δεν είναι δυνατόν γιατί ε, ένα κράτος μέλος τι θα έχει τελικά λόγω του αριθμού των ψηφοφόρων θα είχε μία ή δύο έδρες και κάποιοι άλλοι θα είχαν εκατοντάδες έδρες. Και επομένως είχαμε ένα Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με 5.000 μέλη. 751 ε, ε, έναντι 5.000 καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ μεγάλη διαφορά ήδη και φυσικά Υπάρχουν και διάφορα πράγματα τα οποία θα ήταν ίσως πιο δίκαια, αλλά θα ήταν πολύ δύσκολο και να γίνουν αντιληπτά και να τα δεκτούμε αν μιλήσουμε και με την αρχή ότι μία ε, ψήφος πρέπει να οδηγεί σε μία έδρα. Ε, και ο βασικός στόχος της μεταρρύθμισης θα πρέπει να είναι να, περισσέτει, ε, επιτρέπει περισσότερο στους ψηφοφόρους να έχουν αντίστοιχη εκπροσώπηση με αυτό που ψηφίζουν σε επίπεδο κομμάτων. Τώρα, υπάρχει μια κλασική ε, λειτουργία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η αναλογική ε, ψήφος νομίζω ότι βρίσκεται στις καταβολές αυτού του θέματος. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο φαίνεται σαν ένας χώρος στον οποίο ο, διάφορες πολιτικές δυνάμεις έχουν το λόγο. Αυτό είναι πιο σαφές εδώ και λιγότερο ε, ξεκάθαρο στο Συμβούλιο Υπουργών που έχουμε τις κυβερνήσεις. Η εκλογές θα πρέ... μας επιτρέπουν να έχουμε κάποιες πλειοψηφίες και εδώ είμαστε σε μια πιο κυβερνητική δομή και νομίζω ότι αυτή είναι και μια λογική η οποία ενισχύει και τη ε, διαδικασία του candidate για την επιλογή του Πρόεδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και υπάρχει μια μεταβλητή γεωμετρία. Δεν ναι. υπάρχει μια λογική υποστήριξη ε, μια κυβέρνηση, αλλά υπάρχει ένα συνασπισμό που υποστηρίζει τελικά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και αυτό φυσικά φαίνεται ανάλογα με τα θέματα τα οποία συζητούνται από εκεί και πέρα. Το 70% των ψήφων ε, ε, στις προηγούμενες υποστήριξε μια πολύ μεγάλη, ένα πολύ μεγάλο συνασπισμό. Ε, και από εκεί και πέρα είχαμε ε, συγκεκριμένες ψήφου που πήγανε στην κεντροαριστερά και στην κεντροδεξιά. Και θα υπάρχουν λοιπόν περισσότερες ψήφοι ε, οι οποίες θα πάνε σε ένα μεγάλο συνασπισμό. Αυτό είναι και η επιθυμία των πολιτών ε, και φτάνουμε σε μια διαδικασία που έχει όμως παρόλα αυτά ένα ελάττωμα. Η εκλογική διαδικασία θα πρέπει να επιτρέπει σε μια δημοκρατία την εναλλαγή. εναλλαγή. Από το 1979 ε, η επιλογή των Ευρωπαίων πολιτών είναι να υπάρχει μια, ένας μεγάλος συνασπισμός ή euh, ένα συνασπισμό ο οποίο να είναι αρκετά μεγάλο ε, με βάση συγκεκριμένων συμφωνιών που κάνουν τα κόμματα μεταξύ του. Αυτό ε, έχει επεξεργαστεί και ο Καρλ Πόπερ στο έργο του. Προφανώς και δεν είναι το ίδιο ένας μεγάλος συνασπισμός με το ΕΛΚ στο 36% των ψήφων ή στο 29% και τους φιλελευθέρους. Αλλά για να υπάρχει σαφήνεια για τους πολίτες, ε, τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα. Ε, και δεν είναι δύσκολο για τις χώρες που έχουν μια ε, πολιτική νοοτροπία ε, δυτή, δηλαδή η αριστερά ή δεξιά, η Γαλλία, η Ισπανία, ακόμα και στις χώρες όμως που έχουν νοοτροπία συνασπισμών, όπως η Γερμανία για παράδειγμα, θα μπορούσαμε ίσως πραγματικά να έχουμε κάποιους μεγάλους συνασπισμούς, αλλά δεν έχουμε ένα σύστημα το οποίο μας επιτρέπει πάντα να έχουμε ένα μεγάλο συνασπισμό. Αυτό που λέω είναι ότι δεν λέω ότι είναι παραφύσιν ο μεγάλος συνασπισμός ε, αριστεράς-δεξιάς. Αν το επιθυμεί ο, ε, επιθυμούν οι ψηφοφόροι, ας γίνει. Και εδώ έρχομαι σε κάποιες προσαρμογές που θα επιτρέπουν να μην γίνεται αυτόματα αυτή η διαδικασία και να μπορέσουμε να έχουμε για τους Ευρωπαίους πολίτες μια δυνατότητα ε, σαφέστερης επιλογής. Και προκειμένου να γίνει αυτό, και εδώ θα επισέλθω στις λεπτομέρειες, θα πρέπει να δεχτούμε το εξής και σας το λέω εδώ, θα πρέπει να δεχτούμε για τις δύο μεγάλες ομάδες, για το ΕΛΚ και τους σοσιαλιστές και δημοκράτες, ότι θα βρίσκονται ε, κάποιες φορές ε, στο συνασπισμό που κερδίζει, αλλά και σε κάποιες φορές στο συνασπισμό που χάνει. Ε, επομένως, αυτή είναι η πολιτική στην πραγματικότητα. Να δεχόμαστε ότι πότε κερδίζουμε, πότε χάνουμε. Τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν προκειμένου να βελτιώσουμε την εκλογική διαδικασία και να έχουμε μια, έναν ομοιόμορφο εκλογικό νόμο, ξεκινώντα βέβαια από τη βασική μου υπόθεση, την οποία θα μπορούσε κάλλιστα κάποιο να την αμφισβητήσει. Δεν έχουμε μία ε, μειούμενη αναλογικότητα, έχουμε μία ε, αυξανόμενη αναλογικότητα. Έχουμε μία αναλογικότητα προκειμένου να γίνεται κατανομή των εδρών μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων. Υπάρχει ε, σε πολλά συστήματα ούτως ή άλλως ε, το ε, σύστημα της πριμοδότησης του πρώτου κόμματος με κάποιες επιπλέον έδρες. Γιατί να μην ισχύει και για τις ευρωεκλογέ. Θα μπορούσαμε να προσπαθήσουμε να πάμε σε αυτό, διορθώ, αλλάζοντας την απόφαση του 2002 ή χρησιμοποιώντας ε, τις λύσεις που έχουμε σε διάφορες χώρες. Ποια είναι τα βασικά σημεία εφαρμογής. Τρία τον αριθμό. Καταρχά θα υπάρχουν διάφορα ερωτηματικά για τη διατήρηση της αρχής αναλογικότητα. αναλογικότητας. Αυτό είναι το άρθρο 1 της απόφασης του 2002 που θα μπορούσαμε ίσω να το συζητήσουμε. Ή θα πάμε στη λογική του speech and candidate ή σε μια πιο κυβερνητική δομή όπω ε, όπως έχουμε εδώ, ε, και νομίζω ότι αυτό ε, δεν είναι κάτι το οποίο είναι επιθυμητό, διότι όπως σας είπα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει ε, να διατηρήσει αυτή τη δυνατότητα που έχει να έχει ένα πολύ μεγάλο αριθμό πολιτικών δυνάμεων. Θέλουμε να έχουμε λοιπόν μία αναλογικότητα με πρημοδότηση στα πρώτα κόμματα και εδώ έχουμε δύο στοιχεία τα οποία θα να εξετάσω. Καταρχάς το μέγεθος της ε, εκλογικής περιφέρειας το οποίο βρίσκεται στο άρθρο 2 της απόφασης του Συμβουλίου του 2002, που δίνει τη δυνατότητα να δημιουργούνται εκλογικές περιφέρειες ή εκλογικοί νομοί που δεν λαμβάνουν υπόψη τους απαραίτητο τον αναλογικό χαρακτήρα του εκλογικού συστήματος. όχι στις χώρες που έχουμε πολύ λίγους ευρωβουλευτές, αλλά εκεί που έχουμε πολλούς ευρωβουλευτές, πώς θα μπορούσαμε να πάμε ίσως σε αυτή την κατεύθυνση, ώστε να είναι αντίστοιχοι οι ευρωεκλογές ε, με ε, ε, οι ευρωβουλευτές, συγγνώμη, με τους ψηφοφόρους τους, διότι είναι πολύ μεγάλο το έλλειμμα αυτή τη στιγμή. Ένας Ευρωπαίος Ευρωβουλευτής εκπροσωπεί πολύ περισσότερους πολίτες από έναν εθνικό βουλευτή. Στις κάτω χώρες, για παράδειγμα, ο εθνικός ε, βουλευτής ε, εκπροσωπεί εξαπλάσιο αριθμό ψηφοφόρων. Στη Δανία είναι 13 φορές περισσότερος. Επομένως είναι πάρα πολύ μεγάλο το έλλειμμα. Το οποίο θα μπορούσε ίσως να αυξηθεί περισσότερο σε πολύ μεγάλες εκλογικές περιφέρειες. Αν έχουμε λοιπόν αυτές τις ε, μακροπεριφερειακές εκλογικές περιπτώσεις και ποιο θα ήταν το αποτέλεσμα αυτής της επιλογής, ότι θα είχαμε κάποιες συνέπειες όσον αφορά την πρόσβαση των πολιτικών δυνάμεων κάποιων πιο δευτερευουσό δυνάμεων ίσως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στη Γαλλία για παράδειγμα τι έγινε. Έγινε μεταρρύθμιση του εκλογικού νόμου και πριν από τη μεταρρύθμιση δημιουργήθηκαν, ε, πριν μάλλον από τις 8 ε, μεγάλες περιφέρειες ε, είχαμε τροτσκιστές και κυνηγούς στο κοινοβούλιο. Δεν έχουμε πια τέτοιους. Πρέπει λοιπόν κάτι να γίνει. Και φυσικά αυτό σε καμία περίπτωση δεν είναι απαγορεύσει τι πολιτικέ δυνάμει, αν γίνουν πολύ, πολύ πιο ισχυρέ να έχουν περισσότερε έδρε. Ε, ε ε, Παραδείγματο χάρη υπήρχαν τρει ε, ε, στο Front National στη Γαλλία, τώρα 24 έδρε. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι χρειάζεται μεγαλύτερη ισχύ και πραγματικά εδώ γίνεται μία επιλογή. Ή θα σεβόμαστε συνολικά τον αναλογικό χαρακτήρα ε, του εκλογικού συστήματος όταν καθορίζουμε τις εκλογικές ε, περιφέρειες ή θα μπορούσαμε να έχουμε κάτι επιπλέον για τον αναλογικό χαρακτήρα του ε, συστήματος να λάβουμε υπόψη και το μέγεθος της εκλογικής περιφέρειας. Τρίτο στοιχείο, να υπάρχει ένα κατώτατο όριο για να εισάγεται κάποιος στη Βουλή. Νομίζω ότι αυτό είναι το άρθρο 2.1 της απόφασης του Συμβουλίου. Ε, έχουμε εδώ περίπου το 50% των κρατών μελών, με μικρό ποσοστό, τα είπε κάποιος από τους προηγούμενους ε, ποιοι έχουν εκατότατο όριο εισαγωγής. Εδώ θα μπορούσαμε να έχουμε κάτι το οποίο θα μπορούσαμε να το εφαρμόσουμε, ε, το μεγαλύτερο αριθμό των χωρών, ξεκινώντας από την αρχή ότι ο στόχος των ευρωεκλογών δεν είναι ένα κόμμα το οποίο έχει 1,5% ψήφων και να παίρνει έναν ευρωβουλευτή, αλλά να μπορέσουμε να έχουμε σαφείς πλειοψηφίες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι οποίες θα μπορούσαν να είναι και ε, πλειοψηφίες, για παράδειγμα, ε, του κέντρου, κέντρου αριστεράς, κέντρου δεξιάς ε, κλπ. Σας δίνω λοιπόν και αυτή την άγουσα. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στο σημείο αυτό, ξεκινώντας από τη διαπίστωση που σας παρουσίασα. Και να σας πω ότι νομίζω ότι αυτή η αναζήτηση της σαφήνειας της ιδεολογικής Τάσει των ψηφοφόρων για να τον έχουμε στον εκλογικό νόμο θα πρέπει να αναζητήσουμε ε, με δύο τρόπους. Ε, μέσω του ρόλου των πολιτικών κομμάτων και των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων, τη χρηματοδότηση που θα έχουν, τη δυνατότητα που θα τους δοθεί να κάνουν ε, προεκλογική εκστρατεία, το δυναμισμό τους, το δυναμισμό των ιδρυτών τους και το Και όλα αυτά θα πρέπει να τα αναζητήσουμε επίσης, αν ξεκινήσουμε με αυτή τη διαδικασία, να επικυρώσουμε τις εκλογές μετά όσα συμβαίνουν και εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν ψηφίζει απλώς μόνο κάποιος για να επιλέξει τους ευρωβουλευτές, αλλά υπάρχουν και κάποια όρια τα οποία είναι διαφορετικά. Υπάρχει το όριο της καθολικής ψηφοφορίας, υπάρχει το όριο των μελών ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, υπάρχει το όριο για τα δύο τρίτα, υπάρχει και, το, και η πλειοψηφία των δύο πέμπτων σε κάποιες περιπτώσεις, των τριών πέμπτων, συγγνώμη, αν θέλετε να ακολουθήσετε αυτή τη λογική, λοιπόν, θα μπορούσατε να ακολουθήσετε και αυτή τη λογική των εσωτερικών κανόνων ψηφοφορίας. Δεν καθορίζονται τα πάντα από τη συνθήκη, κάποια καθορίζονται και από τον κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μπορώ να σας δώσω κάποιες λεπτομέρειες. Και θα πρέπει ε, να έχουμε την ψήφο των Ευρωπαίων ψηφοφόρων. Από εκεί και πέρα θα επιτρέπει να επιτρέπει να δημιουργούνται συνασπισμοί, κάποιες φορές και μεταξύ αριστεράς δεξιάς, αλλά να είναι σαφή τα πράγματα και να υπάρχει μια μεγαλύτερη σαφήνεια για τους ε, ε, ψηφοφόρους. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. like to... Ευχαριστούμε πολύ. Αρχίζει τώρα η συζήτηση. Ο Παύλος πρώτος. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Πολύ χρήσιμη και ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Πρέπει όμως να πω ότι έχω την εντύπωση ότι φεύγουμε πάλι από τα ανθρώπινα. Συζητάμε πράγματα που δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτά στο ευρωπαϊκό συνταγματικό πλαίσιο. Well, this issue, because we have been discussing this. Ο κύριος Νταφ μας είπε σημαντικά πράγματα, αλλά νομίζω ότι όσο ήταν εδώ καταφέραμε να τον πείσουμε για μερικά θέματα. Δεν υπάρχει δηλαδή δυνατότητα αλλαγής της σχέσης του σχετισμού δυνάμεων της εκπροσώπησης κάθε χώρας μέλους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αν δεν αλλάξει ταυτόχρονα και το εκλογικό σύστημα. Διότι θα ήταν αφέλεια να πιστεύουμε ότι μπορούμε να εφαρμόσουμε κάποιο μαγικό μαθηματικό τύπο αν και δεν πρόκειται καθαρά για μαθηματικά. Πρόκειται για πολιτικά και θεσμικά θέματα. Μια, ένας μαθηματικός τύπος μπορεί να μας βοηθήσει, αλλά δεν μπορεί να καθορίσει τα πάντα. Τελικά είναι όλα πολιτικές και θεσμικές αποφάσεις. Και για μένα είναι έκπληξη ότι μπορεί κάποιος να προτείνει αναθεώρηση ή μεταρρύθμιση του εκλογικού συστήματος που να σημαίνει μια πολύ ευαίσθητη λεπτή αλλαγή για την κατανομή των εδρών στο Κοινοβούλιο και να μην λέει τίποτα παράλληλα για το Συμβούλιο ίδια θέση δηλαδή που ακούσαμε και από το συνταγματικό δικαστήριο του Γερμανίας όπου και εγώ και άλλοι είχαμε μιλήσει μπροστά σε εννέα δικαστάς μεταξύ των οποίων και ο πρόεδρος Φορσκούλα. Δεν καταλαβαίνω πώς μπορεί ένας Γερμανός νομομαθής που έχει το σύνταγμά του όπου αναφέρεται ότι τα μικρότερα κρατήδια στην Άνω Βουλή έχουν τρία μέλη και τα μεγαλύτερα έξι να ζητάει μεταρρύθμιση της κάτω βουλής και όχι της άνω που για μας είναι το Συμβούλιο. Είναι κάτι που εμείς δεν μπορούμε να το δεχτούμε. Και όταν λέω εμείς δεν εννοώ φυσικά μόνο τις πολιτικές δυνάμεις που εκπροσωπούνται εδώ μέσα και όχι τα μεγάλα ή μικρά κράτη, αλλά τα μέσα, τα μεσαία κράτη, δηλαδή όλα τα κράτη μεταξύ Λετωνίας και Ρουμανίας. Και μπορώ να σας πω ότι και σήμερα ακόμη θα αρχίσουμε τη συνεδρία της θυμακομματική Ομάδας που είχαμε και στην προηγούμενη θητεία όπου γιατί φοβόμαστε ότι θα ξαναρχίσει ο εφιάλτης. Εγώ μπορώ να δεχτώ. Αν είμαστε σε ένα σύστημα που δεν είναι ομοσπονδιακό, πώς μπορούμε να δεχτούμε εκπροσώπηση στην κάτω βουλή όπου οι χώρες δεν παίζουν κανένα ρόλο και το μόνο που παίζει είναι ο πληθυσμός και η δημογραφία τους και απ' την άλλη ένα συμβούλιο όπου ισχύουν άλλοι κανόνες, όχι η ποιότητα, η ποιότητα ενός κράτους. Στην Ελβετία, στις Ηνωμένε Πολιτείες η αρχή είναι ένα κρατήδιο, μία ψήφωση, δύο ή τρεις στην Άνω Βουλή. Δεν ζητάω το ίδιο. Ζητάω τη γερμανική λύση που δεν είναι και πολύ ριζοσπαστική η Πορτογαλία και η Ελλάδα να έχουν τέσσερις ψήφους και οι μεγαλύτερες χώρες έξι. Αν αυτό είναι καλό για τη Γερμανία δεν μπορεί να είναι κακό για την Ευρώπη. Αποκλείεται. Αυτό προσπάθησα να εξηγήσω στον κύριο Φωσκούλα. Αλλά δεν το δεχόταν, δεν το δεχόταν. Θα ήθελα λοιπόν να τονίσω ότι επειδή διδάσκω στη χώρα μου αυτά τα πράγματα συνταγματικό δίκαιο πιστεύω ότι ακούστηκαν εδώ πολλά σοβαρά πράγματα αλλά συνταγματικά και πολιτικά για τις μέσου μεγέθους χώρες δεν θα δεχτούμε καμία αλλαγή Αυτή της εκπροσώπησης εάν δεν συνοδεύεται από πραγματική αλογή στο Συμβούλιο. Και αυτό ισχύει μέχρι την τελευταία μέρα της θητείας μας. Σας διαβεβαιώνω. Έχει ξαναγίνει. Στην έκθεση DAF υπάρχει μια σύνδεση μεταξύ μεταρρύθμισης του εκλογικού νόμου για το Κοινοβούλιο και μεταρρύθμισης του συστήματος ψηφοφορίας στο Συμβούλιο. Δεν είμαστε κατά της αναλογικότητας ή περισσότερης αναλογικότητας στο Κοινοβούλιο. Εφόσον όμως αλλάξει το σύστημα στο Συμβούλιο. Γιατί για μας υπάρχει συνταγματική θεσμική σύνδεση μεταξύ των δύο οργάνων και χωρίς αυτό δεν μπορούμε να δεχτούμε καμία μεταρρύθμιση. Βέβαια αυτό είναι η δική μου απλώς συμβολή στη συζήτηση. Ευχαριστούμε ο Γιώ Λάινεν. ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ και εγώ για τις παρουσιάσεις που ακούσαμε. Παρατηρούμε πόσο πολύπλευρο είναι αυτό το θέμα, το, ο νομός και πόσες προσεγγίσεις υπάρχουν για να κάνουμε ή να μην κάνουμε κάτι. Ο Πάολο Ραγγέλ ήδη έδειξε πόσο δύσκολη είναι μια τέτοια υπόθεση. Να πω πως και η Ρώμη δεν σε μια μέρα και εδώ πέρα θα πρέπει να πάμε σταδιακά. Ίσως και αυτός να ήταν ένας ε, λόγος αυτός για τον οποίο να αποτύχαμε τελευταία, γιατί ξεκινήσαμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα τα οποία δεν μπορούσαν να περάσουν όλα μαζί. Παρ' όλα αυτά, δεν είναι ικανοποιητική η κατάσταση. Ήδη και στη συνθήκη της Ρώμης ε, αναφέρεται μια ενιαία εκλογική διαδικασία. 60 ε, χρόνια μετά έχουμε ένα μοσαϊκό ένα σύστημα το οποίο δεν ανταποκρίνεται στις σημερινές συνθήκες όσον αφορά τις ε, ευρωεκλογές. Τώρα, μια που ο χρόνος πιεζεί να ρωτήσω εγώ τι συζητάμε, ποια είναι η συζήτηση. Έχουμε δύο επίπεδα. Το ένα είναι η προσέλευση στις εκλογές ναι, θα θέλαμε βεβαίως να υπάρχει μεγαλύτερη συμμετοχή, αλλά βλέπουμε πως ε, ισχύει αυτό από τις δημοτικές μέχρι τις ευρωεκλογές, ότι μειώνεται η συμμετοχή. Και βεβαίως έχουμε το θέμα του ότι πρέπει να γίνουν ευρωπαϊκές οι ευρωεκλογές. Δεν έχουμε ευρωπαϊκές εκλογές, έχουμε 28 εθνικές νομοθεσίες, 28 ε, εθνικά ψηφοδέλτια, δεν είναι ευρωπαϊκές οι εκλογές. Αυτό είναι το θέμα. Παρά το ότι έχουμε εδώ και 30 χρόνια άμεση εκλογή του Ευρωκοινοβουλίου και είχε ε, δίκαιο εδώ πέρα ο κύριος Πούκελσχάιμ όταν λέει πως υπάρχει μια απογοήτευση των εκλογέων. Πάνε σε εκλογές που ξέρουν πως δεν είναι ευρωπαϊκές εκλογές, αλλά στα περισσότερα κράτη-μέλη είναι μια εσωτερική αντιπαράθεση. Με τους εθνικούς εκεί πέρα μόνο μάχους που εντάξει είναι οι βασικές μορφές ε, των εκλογών και όχι οι υποψήφοι ευρωβουλευτές. Ίσως θεωρούν πως έχει πολλές, πολύ λίγες αρμοδιότητες ε, το Ευρωκοινοβούλιο. Αλλά αν δούμε τι κρίνεται εδώ πέρα, είναι αποφασιστικό για τη ζωή των πολιτών, αλλά ο πολίτης δεν το μαθαίνει γιατί δεν υπάρχει συζήτηση για την ευρωπαϊκή διάσταση. Ο Γιούργεν Χάμπερμας ε, έλεγε τι είναι ο πυρήνας των εκλογών, της δημοκρατίας. Είναι το να συζητάνε οι πολίτες για αυτά τα οποία κρίνουν την καθημερινή τους ζωή. Δεν υπάρχει ευρωπαϊκή συζήτηση. Εμείς ε, τέσσερις εβδομάδες πριν τις εκλογές ε, κάνουμε μια συζήτηση, αλλά πάντα ασχολούνται με εθνικές συζητήσεις, κάνα σκάνδαλο εθνικό και τέτοια δεν συζητάνε όντως για την Ευρώπη. Οπότε θα πρέπει να δούμε πώς ακριβώς θα υπάρξει μια ευρωπαϊκή κοινή γνώμη. Και εδώ πέρα η συνθήκη της Λισαφωνίας μας δίνει μια εντολή. Είχαν έρθει όλες οι κυβερνήσεις, όλα τα κοινοβούλια δεν είμαστε πλέον ε, εκπρόσωποι μόνο των λαών των κρατών μελών, αλλά και της Ένωσης. Και εκπροσωπούμε το κοινό καλό. Δεν εκπροσωπούμε μόνο τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Πορτογαλία, σύμφωνα με τη συνθήκη, αλλά και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, αυτή ήταν η θεωρία, εν πάση περιπτώσει. Η πράξη είναι κάπως διαφορετική. Και βεβαίως ψηφίζουμε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως ε, νομοθετικό σώμα το οποίο ψηφίζει το εκτελεστικό. Και βεβαίως ε, αυτό έγινε και με τις ακροάσεις, τα ξέρει ο Άντριο Ντάφ, ε, και μετά εγκρίνουμε το σώμα της Επιτροπής Ενοχή. Δεν υπάρχει λοιπόν κάποιο έλλειμμα δημοκρατίας, κύριε Ολύρη. Ο Τζόρτζιο Ναπολιτάνο, όταν ήταν πρόεδρος εδώ πέρα, έλεγε σε αυτό αυτούς που έλεγαν πως ε, δημοκρατία υπάρχει μόνο στο εθνικό επίπεδο και όχι στο ευρωπαϊκό, έλεγε πως έχουμε ε, ελεύθερη καθολική ψηφοφορία. Οπότε η νομιμοποίηση των ευρωεκλογών είναι αυτή ακριβώς των εθνικών ή περιφερειακών κοινοβουλίων ή των δημοτικών συμβουλίων. Ο πυρήνας νομοποίησης είναι η καθολική πυρηνας νομιμοποιησης ειναι η καθολικη ψηφοφορια Βεβαίω καλό θα ήταν να έχουμε προσέλευση άνω του 50%. Αλλά σε κάποιες χώρες γίνεται. Δεν είναι παντού 20%. Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Γερμανία, Αυστρία πλησιάζουν και ξεπερνά το 50%. Στις δημοτικές εκλογές στην πόλη μου ήταν 23% ε, η προσέλευση. Έτσι γίνονται και στις χώρες μας αυτά. Ε, εντάξει, εμείς, εμάς δεν είναι υποχρεωτική η ψηφοφορία βέβαια. Οπότε, καλή η προσέλευση και η συμμετοχή, αλλά αν κολλήσουμε μόνο σε αυτό, θα πάμε προς τα πίσω. Κάνουμε ένα σάλτο μορτάλε προς τα πίσω. Τα είπε ο κύριος Σολύρη. δεν θα είναι ευρωπαϊκές οι εκλογές και θα οπισθοχωρήσει ο τροχός της ιστορίας προς τα πίσω. Πρέπει να ζητήσουμε ε, στοιχεία για αυτή την ευρωπαϊκή συζήτηση, για ευρωπαϊκά αγαθά, για ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Και θεωρώ πως ήταν μια καλή αρχή το σύστημα αυτό των υποψηφίων. Ε, μέχρι και ο David Cameron αναρωτήθηκε τι είναι αυτή η Spitzenkandidaten δεν ξέρω, θα μπορούσαν ας πούμε, να είναι και στις 28 χώρες. Ε, υπερεθνικές λίστες, ναι, θετικό. Το έχουμε ζητήσει εδώ και 20 χρόνια. Αλλά βεβαίως ε, το θέμα μετά πάει στις συνθήκες και στο πρωτογενές δίκαιο. Δεν ξέρω αν θα γίνει μέχρι το 2019, αλλά πρέπει να παραμείνει η συζήτηση. Η διπλή αναλογικότητα Πράγματι, είναι ενδιαφέρον το σύστημα. Αυτό πρέπει να μας απασχολήσει. Έστω και αν δεν πετύχουμε την ιδανική λύση. Γιατί αντικατοπτρίζει και το διπλό επίπεδο της Ένωσης. Η ταυτότητα της Ένωσης είναι μια διπλή νομοποίηση μέσω των κρατών και των πολιτών και αυτή η διπλή αναλογικότητα αντικατοπτρίζει κάπως το ευρωπαϊκό επίπεδο, το πολιτικό δηλαδή και το εδαφικό στο επίπεδο του κράτους μέλους. Κύριε Πούκελσχάιμ, έχω μια ερώτηση για σας. Γιατί πέρα από τα ευρωπαϊκά κόμματα που έχουμε ήδη χρειαζόμαστε μια νέα κατασκευή Έχουμε 12 ε, οικογένειες κομμάτων από τέρμα δεξιά μέχρι τέρμα αριστερά. Και έχουμε εντάξει αυτή τη, την όθηση που έχουμε να οργανωνόμαστε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Α, εντάξει δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα. Δεν γίνεται να έχουμε και τα αυγά και την ε, ομελέτα. Το να κατεβαίνει κανείς σε ευρωεκλογές σημαίνει πως θα είναι ένας ευρωπαϊκός σχηματισμός. Εντάξει, το 2019 μπορούμε να κάνουμε κάποια πράγματα, να αναφέρονται στο ψηφοδέλτιο τα ευρωπαϊκά κόμματα, ίσως ε, στο εκλογικό υλικό οπωσδήποτε, ένα ελάχιστο κατόφλι πράγματι θα, σε όλες τις χώρες θα δημιουργήσει μια κάποια ισότητα και νομίζω πως κάποια χρήσιμα πράγματα ακούσαμε τα οποία θα συμπεριλάβουμε και ως αύκο στην πρότασή μας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ράινερ Βίλαντ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα, να πω το εξή πως πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τα της Λισαβόνας πριν κάνουμε παραπέρα βήματα. Η σκέψη που ακούσαμε... Εντάξει, καλές είναι, αλλά Δεν ξέρω εάν θα χρειαστεί να αλλάξει τίποτα στον ε, εκλογικό ε, νόμο. Δεν νομίζω να χρειαστεί δηλαδή να αλλάξει τίποτα. Δεύτερον, στο σύνταγμα της δικιάς μου ε, χώρας μιλά, οι εκλογές λέγονται ότι πρέπει να είναι ελεύθερες, καθολικές και μυστικές. Το ελεύθερες δεν είναι ακριβώς ελεύθερες, γιατί στο Βέλγιο είναι υποχρεωτικές, ενώ εγώ μπορεί να αποφασίσω ότι δεν θέλω να πάω, να ψηφίσω. Και βεβαίως το ουσιαστικό είναι το εάν είναι ε, ίση η ψήφος του καθενός. Και εγώ δεν θεωρώ τώρα για ένα άλλο θέμα δεν θεωρώ ότι πρέπει να συζητάμε καν το θέμα της προσέλευσης της ευρωεκλογές. Αυτό συμβαίνει παντού. Έχω εδώ πέρα ένα έντυπο από την υπηρεσία του Κοινοβουλίου που δείχνει πως η προσέλευση των ευρωπαϊκών ε, εκλογών κινείται ακριβώς παράλληλα με την προσέλευση στις ε, εκλογές στην Αμερική για το Κογκρέσο και τον Πρόεδρο. τα τελευταία 30 χρόνια. Εντάξει, ναι, να προσπαθήσουμε για μεγαλύτερη προσέλευση, αλλά δεν σημαίνει αυτό ότι με λιγότερη ή περισσότερη προσέλευση έχουμε λιγότερη ή περισσότερη νομοποίηση. Θα είπε και ο κύριος Λάινεν. Αυτά γίνονται και στους δημάρχους, στις δημοτικές εκλογές. Και τα τελευταία 5, 50 χρόνια βλέπουμε αυτή την εξέλιξη. Συν το ότι έχουμε χώρες που εντάσσονται, βλέπετε την ε, Κροατία που έχει πάρα πολύ χαμηλά ε, ποσοστά συμμετοχής. Και γενικά ε, οι χώρες οι οποίες προσθέθηκαν πιο πρόσφατα το παρουσιάζουν αυτό το φαινόμενο. Μπορείτε να δείτε αυτό εδώ πέρα, το, το έγγραφο είναι χαρακτηριστικό. Κατόπιν, υπερεθνικές λίστες. Ωραία η ιδέα. Ε, είπε ο κύριος Λάινεν να πάμε σιγά σιγά. Ναι εντάξει αλλά ας σκεφτούμε ότι χτίζουμε ένα κτίριο ξέρω εγώ μια εκκλησία οι υπερεθνικές λίστες είναι το καμπαναριό έτσι είναι το, το τελευταίο το είπε και ο κύριος ε, Πούκελσχάιμ ότι τα τρία τέταρτα θα ήθελαν εθνικές λίστες. Μα, δηλαδή, θεωρείτε πραγματικά ότι αν πλακοθούμε εδώ πέρα με τον συνάδελφο Ράγκελ, πλακοθούμε για μία έδρα παραπάνω, έχει κάποιο νόημα αυτή η συζήτηση για το αν θα έχουμε ένα Μαλτέζο παραπάνω. Εντάξει, μην προσβάλλουμε και την νοημοσύνη μας. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, τι ξέρω, θα γίνει πάρα πολύ δύσκολα. Πάντα το λέμε, το αναφέρουμε στα εκτιμώντας, αλλά είναι κάτι το οποίο θα γίνει πάρα πολύ δύσκολα. Ήδη τα είδαμε αυτά και πέρσι και ποιο ήταν το αποτέλεσμα. Δεν πήραμε τίποτα άλλο από αυτά τα οποία θέλαμε, γι' αυτό μείναμε με τις ε, υπερσμικές λίστες ως ζητούμενο. Μετά, δημοκρατικό έλλειμμα. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε στο Γερμανικό Συνταγματικό Δικαστήριο να ξαναμιλήσει για δημοκρατικό έλλειμμα. Και κύριε Ράγγελ, Δεν μπορεί να πούμε μετά, α, ναι, τότε θα κάνουμε το γερμανικό σύστημα. Γιατί, γιατί το γερμανικό σύστημα, τι σημαίνει, ότι στην Κομισιόν, την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση δηλαδή, δεν θα εκπροσωπείται κάθε χώρα. Δεν μπορούμε να διαλέγουμε όσα μας αρέσουν μόνο από ένα σύστημα, γιατί εδώ πέρα στην ε, Κομισιόν έχουμε έναν αναχώρα, στο Συμβούλιο έχουμε μια διπλή πλειοψηφία, δηλαδή έχουμε και δύναμη αλλά και αναχώρα και στο Κοινοβούλιο ψάχνουμε μια άλλη μέθοδο. Τι να σας πω. Δεν θα ξεφύγουμε από τον ε, εφιάλτη στην επόμενη διεύρυνση ή μετά από αυτήν θα έχουμε ξανά την ίδια αυτή συζήτηση. Εάν δεν καταλήξουμε σε μία ε, λύση. Κύριε Νταφ, κύριε Πούκελσχάιν, όταν μιλάμε συγκεκριμένα για μια συνταγή, εάν θέλετε, ή για μια λύση, πρέπει πάλι και με την προτινόμενη λύση θα ε, έχουμε το εξής πρόβλημα. Αν δεν μπορούν οι δάσκαλοι να εξηγήσουν στους μαθητές πώς εκλέγεται το κοινοβούλιο, έχουμε πραγματικά πρόβλημα. Και αυτό ισχύει νομίζω για τον συμβασμό του Κέμπριτς που έχετε προτείνει. Γιατί δύο τρίτα των Ευρωπαίων πολιτών ψηφίζουν σε κλειστές λίστες. Αυτό θεωρούν δηλαδή τα δύο τρίτα των πολιτών ε, δημοκρατία. Και, στα, και επίσης το σύστημα DEONT, ανεξαρτήτως του πώς το ονομάζουν. Πρέπει λοιπόν να μπορούμε να τα εξηγήσουμε αυτά στον κόσμο. Δεν ζούμε μόνο στο, στο δικό μας τον κλειστό κόσμο. Και για να μην έχουμε συνέχεια την ίδια συζήτηση, τα θυμάμαι και στο παρελθόν, σε κάθε διεύρυνση. Γιατί τελικά τι έγινε, ο καθένας ε, εξασφάλισε τους δικούς του και έμεινε τελευταία η Αυστρία με τη Σουηδία να ε, την πληρώσουν. Κόμματα τώρα. Δεν πρέπει τώρα να προκαθορίσουμε εμεί τι μέγεθος θα έχει το, το σηματάκι πάνω στο ψηφοδέλτιο ή τη γραμματοσυρά και μέγεθος. Ε, για το όνομα του Θεού. Α τα κάνει αυτά η κάθε χώρα, ο κάθε νομοθέτης ανάλογα με το δικό του εκλογικό νόμο. Όποιο κόμμα θέλει να, να βάλει από πάνω το Ευρωπαϊκό Κόμμα και τον Ευρωπαίο Υποψήφιο το κάνει. Αυτό φτάνει. Όσοι θέλουν το κάνουν, όσοι δεν θέλουν δεν το κάνουν. Αλλά όσοι θέλουν να μπορούν. Αυτό φτάνει. Αυτό για μένα φτάνει. Τώρα το τι μορφή θα έχει ακριβώς το ψηφοδέλτιο, ας μην κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Και να μην περάσουμε πάλι ξανά σε συζήτηση για την ε, ηλικία, που είναι πάλι μεγάλο θέμα στην ε, Γερμανία. Δηλαδή τέτοιες σοβαρές αλλαγές ε, στο αστικό δίκαιο της κάθε χώρας ε, δεν μπορεί να τις ε, κάνουμε έτσι χωρίς να σκεφτούμε. Ή ε, ας πούμε ξέρω εγώ κάτι, μια κλίμακα από 16 έως 21 και άμα κινείσαι εκεί μέσα, καλώς. Επίσης κάτι άλλο που δεν το ανέφερε κανένας ειδικός. θέλουμε μια ευρωπαϊκή δημοκρατία με ελεύθερες εκλογές κτλ. Και, και πόσο λίγο έχουμε ασχοληθεί με το πόσο δημοκρατικά επιλέγονται οι υποψήφοι στις χώρες. Δεν το αναφέρει απολύτως κανένας. Υπάρχουν χώρες που, ε, στις οποίες το κόμμα ή ο πρόεδρος του κόμματος ετοιμάζει τη λίστα ή πολύ μικρά σώματα Υπάρχουν χώρες που η λίστα εμφανίζεται 10 μέρες πριν τις εκλογές. Δεν είναι δυνατόν να γίνεται κάτι τέτοιο. Για μένα η χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών κομμάτων πρέπει να εξαρτηθεί από την εσωκομματική δημοκρατία. Ή τουλάχιστον στο πώς επιλέγονται οι υποψήφοι. Και μετά από εκεί και πέρα βλέπουμε. Έτσι. Αλλά αυτό πρέπει να είναι βάση. Ο μεγάλος συνασπισμός τώρα. Εντάξει, πρέπει να μου αρέσει, αλλά δεν μπορεί να λέμε τη μία μέρα να λέμε θέλω πλειοψηφία την άλλη μέρα να, θέμε, να λέμε θέλω μεγάλο συνασπισμό ανάλογα με τα γούστα. δούμε ποιες από αυτές τις δυνατότητες θα ακολουθήσουμε. Εντάξει, οι υποψήφοι αυτοί ήταν νομίζω μία επιτυχής ε, ιδέα. Και ας αναρωτιέται ο κύριος ε, Κάμερον. Στη χώρα μου στη, και στο δικό μου το κρατήδιο τι να σας πω, ήταν υποψήφιο ο κύριος Στάινμαερ και η κυρία Μέρκελ. Δεν εμφανίστηκαν στο κρατηδιό μου παρόλα αυτά. Δεν είναι κανένα συνταγματικό πραξικόπημα αυτό το πράγμα. Και εδώ πέρα στη δικιά μας την περίπτωση δεν έχουν λόγο οι αρχηγοί των κυβερνήσεων, έχουν λόγο οι αρχηγοί των κομμάτων, τα μέλη των κομμάτων και λένε αυτός είναι ο δικός μας ο υποψήφιος. Αυτό το κάνουν τα κόμματα, όχι οι αρχηγοί των κυβερνήσεων. Δεν μιλάω για την ταυτότητα έτσι, των προσώπων, αλλά και για το τι θα κάνουν. Έτσι, και δεν χρειάζεται τίποτα να αλλάξει εδώ πέρα νομοθετικά και στη Γερμανία ε, η έννοια αυτή του υποψηφίου του κάθε κόμματος δεν υπάρχει σε κανένα νόμο, ούτε στο Σύνταγμα, ούτε πουθενά. Μην μπερδεύουμε τη, τις διαφορές με τα πρόσωπα και το τι φαίνεται στα μημύε. Κάτι άλλο που είναι σημαντικό για μένα το θέμα του κατακαιρματισμού του Κοινοβουλίου. Και εδώ πέρα μπορούμε να δούμε λίγο τους αριθμούς. Μια χώρα που έχει 10 βουλευτές και ένα ας πούμε κανονικό εκλογικό δίκαιο έχει de facto έτσι, ένα κατόφλι 10%. Εντάξει, στα, στα άκρα βεβαίως, ε, στα μαθηματικά πάντα διαφέρουν τα πράγματα, αλλά κατά κανόνα μια χώρα που έχει 10 βουλευτές, ποιο είναι το όριο για να βγάλεις ένα βουλευτή, 10%. Και ο κατακαιρματισμός του Κοινοβουλίου όμως δεν γίνεται από την Κύπρο, ούτε από τη Μάλτα. Από τις μεγαλύτερες χώρες προκύπτει. Γι' αυτό υπάρχει κάποια λογική ε, όταν λέμε πως ε, οι χώρες που είναι ξέρω, πάνω από 10 εκατομμύρια, πάνω από το 2% του πληθυσμού, υπάρχει το όριο του 5%. Εκεί πέρα να πούμε ότι έχουμε ένα όριο 5 ή 4%. Οπότε μπορούν οι Ιρλανδοί να παραμείνουν στο σύστημά τους και να μην έχουμε κανένα πρόβλημα και αποφεύγουμε και τον καταγρηματισμό του Κοινοβουλίου και πάμε σε μια, σε αυτή την καινοτομία. Τι όλα τα υπόλοιπα, ε, εγώ είμαι κάπως επιφυλακτικός. Εντάξει, είμαι πεπισμένο ότι χρειάζεται μια άλλη λύση, αλλά δεν ξέρω αν θα την επιτύχουμε στο τέλο. Γιατί και οι υπόλοιποι Γερμανοί συναδελφοί μου μου λένε πω ε, βλέπουμε πω πάμε σε ε, ένα αμάλγαμα. Δηλαδή, ε, να έχουμε μια βάση και θα λέμε κάθε χώρα θα έχει τόσους βουλευτές και το υπόλοιπο ανάλογα με το σύστημα DEONT. Με το ανώτατο όριο που υπάρχει βεβαίως. Κάτι το οποίο καταλήγει σε πολύ παρόμοια αποτελέσματα με τον συμβιβασμό του Κέμπριτς και, ξαναλέω, μπορεί να το εξηγήσει ο δάσκαλος σε ένα σχολείο. Ε, thank you very much, George. Ευχαριστούμε πολύ. Ο Νταφ. Όχι, ο Τζόρτζ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η συζήτηση μέχρι τώρα ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και θα ήθελα να θίξω μερικά θέματα με βάση αυτά που είπαν και άλλοι. Πρώτον, το όλο θέμα των υπερεθνικών ψηφοδελτίων. Εσείς τις λέτε πανευρωπαϊκές, αλλά βέβαια δεν είναι αυτό. Όταν ήμουν ο σκιώδης σου, Ανδρέα, Ήμουν μετρίος υπέρ, αλλά οι συζητήσει στο ΕΛΚ μου με όθησαν προς κάποιες περισσότερες αμφιβολίε. Ενώ ο συμβιβασμό του Κέμπριτζ, στη σελίδα 12 του εγγράφου του Ανδρέα, βλέπετε ότι η χώρα μου η Ουγγαρία είναι πολύ χρήσιμο παράδειγμα. Μπορείτε να φανταστείτε να πω στους συμπολίτες μου θα χάσουμε τέσσερις ευρωβουλευτές με βάση αυτό το σχέδιο, τέσσερις έντρες. Έπειτα, τα στατιστικά στοιχεία λένε ότι οι Ούγγροι είναι λίγο κάτω από 10 εκατομμύρια, αλλά ο αριθμός των Ούγγρων πολιτών στην Ευρώπη είναι ίσως 10 και μισό εκατομμύρια. Έχουμε πολλούς Ούγγρους δηλαδή που ζουν σε άλλες χώρες και που δεν εκπροσωπούνται. Μπορούμε σοβαρά να πούμε ότι ένας ε, βουλευτής του UKIP θα εκπροσωπεί και Ούγγρους και Ρουμάνους ή ότι το Ποδέμος θα εκπροσωπεί και Βρετανούς συνταξιούχους που ζουν στην Ισπανία. Δεν συμβαίνουν αυτά. Ίσως 8 με 10 εκατομμύρια Ευρωπαίοι να μην εκπροσωπούνται επαρκώς στο Κοινοβούλιο. Καλός ο συμβιβασμός του Κέμπριτζ, αλλά νομίζω ότι δημιουργεί και μία εκλογική αδικία. Οι μικρομεσαίες χώρες δεν πρόκειται να τη δεχτούν. Όσο για τις κινήσεις των πληθυσμών δεν θα σταματήσουν αυτά, είναι μια δυναμική διαδικασία και πρέπει να προσαρμοστεί σε αυτήν τη λύση του Κέμπριτζ για να τη δεχτούν και οι πολίτες. Έπειτα. Μπόκουσχάιμ μίλησε για παραπλάνηση του εκλογικού σώματος, αλλά θα μπορούσαμε να το δούμε και αλλιώς. Υπάρχει πολύ λίγη ταύτιση του πολίτη με την ε, άσκηση των δικαιοδοσιών των Ευρωβουλευτών. Ίσως θυμάστε τι έγινε με το δεύτερο Ιρλανδικό δημοψήφισμα. Ο κόσμος δεν μπορεί, καλός ή κακός, να ταυτίσει τους Ευρωπαίους πολιτικούς με τους δικούς του. Τι είναι αυτή η Ευρώπη, κανείς δεν ξέρει, είναι η πολυπλοκότητα των θεσμών για την οποία μίλησε και ο Ανδρέας. Είναι όντως πολύ δύσκολο να ταυτιστεί κανείς με το ευρωπαϊκό επίπεδο πολιτικής. Εμείς εδώ το κάνουμε, αλλά ακόμη και για μας χρειάζεται αρκετός χρόνος για να καταλάβουμε περί τίνος πρόκειται, γιατί είναι πολύπλοκα όλα αυτά. Μόλις φτάσουμε δεν ξέρουμε ήδη πώς λειτουργούν τα πράγματα και μου φαίνεται ότι για τον περισσότερο κόσμο η πολιτική είναι κάτι εθνικό και τις ευρωεκλογέ έτσι τις βλέπουν εθνικά. Εγώ μπορεί να λέω αυτά που γίνονται στην Ευρώπη, αλλά ο κόσμος απαντάει εντάξει πολύ ενδιαφέρον αυτό, αλλά πώς θα κερδίσουμε τους σοσιαλιστές. Αλλάζει λοιπόν η συζήτηση αμέσως. Το θέμα είναι λοιπόν πώς θα εκλαϊκευτεί, θα περάσει στον κόσμο αυτή η έννοια του ευρωπαϊκού κοινού αγαθού. Η ελίτ ίσως τα καταλαβαίνει αυτά, αλλά δεν έχουν φτάσει στον κόσμο. Δεν λέω ότι έχουμε αποτύχει, αλλά δεν έχει ακόμα φτάσει. Τρίτον, η προφανής μείωση, αύξηση μάλλον της αποχής. Το είπε και ο Βίλαντ. Οι περισσότερες, στις περισσότερες σύγχρονες δημοκρατίες δεν είναι υποχρεωτική η ψήφος. Υπάρχει η αποχή, το ευδιευκολύνει αυτό, αλλά υπάρχει και μια άλλη εξήγηση. Η εξουσία στις σύγχρονες δημοκρατίες έχει ανακατεμινεμηθεί. Πριν από 50 χρόνια οι νομοθέτες ασκούσαν την εξουσία. Τώρα όχι πια. Έχουν, έχει δοθεί και σε λόμπι και σε μη κυβερνητικέ οργανώσεις και στους δικαστάς. Και το αποτέλεσμα είναι ότι για πολλούς λόγους από λέει ότι δεν τον ενδιαφέρουν οι ευρωεκλογέ. Ο κόσμος είναι λογικός. Μερικοί μπορεί να έχουν συγκεκριμένα προβλήματα που δεν λύνονται από το ευρωπαϊκό επίπεδο κτλ. Και επομένως μειώνεται η συμμετοχή και αυτό είναι χαρακτηριστικό της σύγχρονης δημοκρατίας, είτε μας αρέσει είτε όχι. Τέλος, αν περάσουμε στην προοδευτική αναλογικότητα, αυτό θα ενισχύσει την ανακατανομή των εξουσιών στο Κοινοβούλιο που πρέπει να το σκεφτούμε σοβαρά, αλλά επίσης και τις δικαιοδοσίες των μεγάλων χωρών μελών και οι μικρότερες θα ανησυχήσουν. Εγώ δεν είμαι βέβαιος σε τι βαθμό οι μεγαλύτερες χώρες μέλη είναι διατεθειμένες να εφαρμόσουν τη δημοκρατική αρχή του αυτοπεριορισμού. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα νομίζω. Και επομένως, όποιες και να είναι οι ατέλειες του υπάρχοντος συστήματος, είναι καλύτερο για τις μικρομεσαίες χώρες, εκπροσωπούνται καλύτερα, γιατί γενικά έχουν εθνικά συμφέροντα και ευρωπαϊκά, συμμετέχουν στο ευρωπαϊκό επίπεδο και δεν πρέπει να παραγνωριστούν αυτά υπέρ των συμφερόντων των μεγάλων κρατών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριος Κατρούγκαλος. Thank you, Mr. Chair. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Η πρώτη μου παρατήρηση είναι ότι δεν είναι δυνατόν να δώσουμε λύσεις σε πολιτικά προβλήματα μόνο μέσω τεχνικών οδών. Και το ολοκληρωτικό σύστημα είναι σαφώς ένα τεχνικό μέσο. Ποιο είναι το βασικό πρόβλημα της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας. Ακούσαμε ήδη δύο συμπτώματα. Πρώτον, από τον καθηγητή Νταλιμόντε, ότι για το μέσο πολίτη οι εκλογές φαίνεται ότι δεν έχουν καμία σημασία για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δεν είναι αποφασιστική σημασία. Και τώρα ο συνάδελφος ο Τζορτ Σόπφιλ μόλις μας είπε ότι γι' αυτό το λόγο ψηφίζουμε ακόμα και στις ευρωπαϊκές εκλογές με εθνικά κριτήρια. Και γιατί συμβαίνει αυτό νομίζω ότι η απάντηση είναι προφανής. Στην Ευρώπη δεν υπάρχει ένας κοινό ευρωπαϊκός δημόσιος χώρος. Και αυτό διαφέρει από την ύπαρξη μιας ευρωπαϊκής πολιτείας. Δεν είναι εύκολο να έχουμε στο ε, εγγύς μέλλον ε, μια ευρωπαϊκή πολιτεία και δεν νομίζω ότι είναι και ε, επιθυμητό αυτό. Από την άλλη είναι επιβεβλημένο να υπάρχει ένας κοινό ευρωπαϊκός χώρος υπό την έννοια ότι θα έχουμε και τη δυνατότητα να συζητήσουμε τα πιο σημαντικά πολιτικά ζητήματα οριζόντια σε όλα τα κράτη-μέλη με το ίδιο πολιτικό θεματολόγιο. Η αρχή της δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού δημοσίου χώρου ίσως να μας επιτρέπεται μέσω της υπόθεσης του Spitzenkandidat. Δηλαδή, παρουσιάστηκαν σε όλο το Ευρωπαϊκό Εκλογικό Σώμα με κάποιο συγκεκριμένο πολιτικό θεματολόγιο το οποίο ήταν το ε, ε, πρόγραμμα του πολιτικού του κόμματος. Αλλά κατά την άποψή μου το θέμα δεν είναι μόνο αυτό. Το θέμα είναι να υπάρξει και κατανόηση και να ε, γίνει δεκτό ότι κάποια κρίσιμη σημασία πολιτικά ζητήματα είναι θέμα κοινού ενδιαφέροντο για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παραδείγματο χάρη η ενίσχυση της πρωτοβουλία των πολιτών και τη σχετική ρήτρα. Εάν μπορούμε να έχουμε ένα δημοψήφισμα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο για κάποιο κρίσιμο ζήτημα, αυτό θα δημιουργούσε μια πολύ διαφορετική προσέγγιση από την προσέγγιση που είχαμε στα δημοψηφίσματα που σχετίζονταν με την επικύρωση των συνθήκων. Διότι ακόμα και τα συγκεκριμένα δημοψηφίσματα και ε, ε, ε, απάντηση είχαν άμεση σχέση με τις εσωτερικές πολιτικές. Αντιθέτως, εάν υπάρχει μια γενικευμένη συζήτηση για ένα θέμα μεμονωμένο, θα μπορούσε για παράδειγμα να είναι η λιτότητα ένα εξ αυτών, θεωρώ ότι αυτό θα μπορούσε να συνεισφέρει πραγματικά στην ε, ε, δημιουργία αυτού του ευρωπαϊκού χώρου. Τελευταία παρατήρηση, η μικρή συμμετοχή είναι ένδειξη ε, σχετικής απώλειας ευρωπαϊκής νομιμοποίησης. Και νομίζω ότι δεν θα πρέπει να συγκρίνουμε τη συμμετοχή στις ευρωεκλογέ με τη συμμετοχή στις Ηνωμένε Πολιτείες διότι αναφερόμαστε σε μια τελείως διαφορετική πολιτική νοοτροπία. Νομίζω ότι η μόνη λογική σύγκριση θα ήταν να τις συγκρίνουμε με τη συμμετοχή ε, στις εκλογές στα εθνικά κοινοβούλια, για τα εθνικά κοινοβούλια. Και εκεί νομίζω ότι είναι σαφές ε, το θέμα της διαφοράς. Είναι πολύ σοβαρή διαφορά που υπάρχει. Και τέλος, όσον αφορά το θέμα της νομιμοποίησης, θεωρώ ότι είναι σαφής ο λόγος για τον οποίο υπάρχει. Ποιο ήταν ο βασικός τρόπος νομιμοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο καθηγητής Βάιλερ μας είπε σαφέστατα ότι ήταν ε, μία νομιμοποίηση η οποία είχε ε, προέλθει προς τα έξω η Ευρωπαϊκή Ένωση αφορούσε όλα τα κράτη-μέλη και ο Ευρωπαίος πολίτης θεωρούσε ότι το ευρωπαϊκό όραμα είναι κάτι το οποίο βελτιώνει την προσωπική του ζωή, την προσωπική του κατάσταση. Αν το είχαμε δεχτεί ως έτσι, ε, δεν θα υπήρχε πρόβλημα, ακόμα και αν ξεκινούσε προς τα κάτω ευθύς εξ αρχής. Όταν αυτό εξαφανίστηκε με την εφαρμογή των πολιτικών λιτότητας, είναι σαφές ότι δεν μπορεί πλέον να υπάρξει ε, σωστό το σύστημα. Και θεωρώ λοιπόν ότι πέραν του διαρθρωτικού προβλήματος, που είναι η ανυπαρξία του ευρωπαϊκού ε, δημοσίου χώρου, ο πολύ σημαντικός ε, λόγος για την κρίση της νομιμοποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι οι πολιτικές αυτές. Ευχαριστώ, Γιώργο Ρίτσαρτ Κόρμπετ. Ευχαριστώ. Μου άρεσαν πάρα πολύ οι παρουσιάσεις, ε, προσφέρουν τροφή για σκέψη. Αλλά ως προς το πώς θα ανταποκριθούμε εμεί τώρα ως ε, Επιτροπή Σταγματικών Υποθέσεων και ως Ευρωβουλευτές, νομίζω ότι θα πρέπει να εξετάσουμε πάρα πολύ προσεκτικά τι μπορούμε να αλλάξουμε και τι έχει πραγματικά σημασία. Εξάλλου, είμαστε ένα μέσο στο οποίο συνταγματικέ αλλαγέ, όταν λέω συνταγματικέ αλλαγέ, εννοώ ουσιαστική αλλαγή των κανόνων μα, των εθνικών μα, οι συνταγματικέ αλλαγέ αποτελούν ε, αντικείμενο ομοφωνίας από τα κράτη-μέλη και εθνική επικύρωση. Και κάποια από τα θέματα που συζητήσαμε σήμερα προϋποθέτουν συνταγματικές αλλαγές και κάποια από αυτά νομίζω ε, ότι έχουν ελάχιστες πιθανότητες να συμβούν. Όταν λοιπόν θα προχωρήσουμε τις εργασίες μας, θα πρέπει καταρχάς να εξετάσουμε ποιο είναι πραγματικά το πρόβλημα, παραδείγματο χάρη, το γεγονό ότι υπάρχουν διαφορετικά όρια ηλικία για να συμμετέχει κάποιο ω υποψήφιο σε εκλογέ στα κράτη-μέλη, είναι πραγματικά πρόβλημα για το σύστημα, για εμά ω Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ω Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν νομίζω. Είναι κάτι το οποίο ε, μπορούμε να δεχτούμε, διότι. Ε, σύνθημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ε, συνυπάρχουμε μέσα από τη διαφορετικότητα. Το γεγονός ότι άλλοι χρησιμοποιούν ε, σύστημα αναλογικό don't και άλλο, ένα άλλο αναλογικό σύστημα, δεν ξέρω. Το να χρησιμοποιούν κάποιοι διπλή αναλογικότητα, δεν ξέρω αν είναι πρόβλημα, ίσως είναι, αλλά και αυτό μπορούμε να το αντέξουμε. υπάρχουν κάποια πράγματα οποία ίσως θα επιθυμούσαμε να αλλάξουμε, αλλά οι πιθανότητες να αλλάξουν είναι πάρα πολύ ισχνές. Παραδείγματος χάρη, το να περάσουμε στην απλή αναλογικότητα για την κατανομή των εδρών μεταξύ των κρατών μελών. Καμία περίπτωση να υπάρξει συμφωνία. Κάτι το οποίο ίσως ε, θεωρούμε υπερβολικά ε, πρόβλημα. Εγώ προέρχομαι από το Ηνωμένο Βασίλειο όπου έχουμε Σκοτσέζους, Ουαλούς, ε, τη Βόρεια Ιρλανδία και έχει πολύ μεγαλύτερη εκπροσώπηση από αυτούς σε σχέση με την Αγγλία. Αυτό δεν είναι αναλογικό, είναι μεγάλο πρόβλημα. Δεν είναι μεγάλο πρόβλημα, υπάρχουν κάποια άλλα προβλήματα αλλά όχι αυτό. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ε, μπορούμε να ζήσουμε και με αυτό. Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι ίσως είναι πάρα πολύ μεγάλο. Um, το να φτάσουμε μέχρι ή και τέσσερις τέλος πάντων να δεχτούμε τους πέντε τώρα. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο αποτελεί πρόκληση για το όλο σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και Παρεμπιπτόντως, όλοι αυτοί οι παράγοντες δεν ε, καθορίζουν το ποσοστό συμμετοχής στις εκλογές κατά την άποψή μου. Ίσως ε, κάποιο ε, περιθώριο, κάποιο μικρό ποσοστό αλλαγής, αλλά όχι το σύνολο. Και όσον αφορά το ποσοστό συμμετοχής, όταν λέω γι' αυτό. Θα ίσως πρέπει να το αναλύσουμε λίγο περισσότερο και να εξετάσουμε την τάση και το επίπεδο. Νομίζω ότι είναι λογικό ότι οι ευρωεκλογέ έχουν χαμηλότερο επίπεδο συμμετοχής από τις εθνικέ εκλογές. Άλλωστε, είναι όσα έχουν αυτή τη στιγμή λιγότερο σημαντικέ και παρεπιπτόντω δεν διακυβέρνεται η κυβέρνηση. Οι περισσότεροι άνθρωποι όταν ψηφίζουν στι εθνικέ εκλογέ, επιλέγουν αν θα διατηρήσουμε αυτή την κυβέρνηση ή θα την αλλάξουμε. Αυτό είναι το ναι. κίνητρο των ανθρώπων και αυτό φυσικά δεν προβάλλεται με αυτόν τον τρόπο στι ευρωεκλογέ. Ε, αρχίζει να γίνεται ίσω με του ε, speech candidates, του επικεφαλεί για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά αν αρχίσει αυτό το σύστημα να λειτουργεί λίγο καλύτερα, τότε ίσω θα έχουμε κάποιες πιο ουσιαστικές αλλαγές σε επίπεδο συμμετοχής στις εκλογές. Και παρεμπιπτόντως αυτό είναι και κάτι το οποίο δεν απαιτεί αλλαγή της συνθήκης. Όπως ήδη επισημάνθηκε, επαφίεται στα πολιτικά κόμματα στον τρόπο με τον οποίο ε, θα ε, ε, συνεργαστούμε την κοινή γνώμη και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης θα μπορούσε να αποτελέσει και αυτό ένα απόσπαστο τμήμα της εκλογικής διαδικασίας και να θεωρήσω ο ψηφοφόρος ότι η ψήφος μου είναι συνιστόσα του πώς θα ηγείται τουλάχιστον ε, κάποιος του εκτελεστικού οργάνου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, ε, διότι το άλλο θα είναι ούτως ή άλλως ένα συνασπισμός. Δεν μπορεί να αλλάξει αυτό χωρίς να αλλάξουν οι συνθήκες, αλλά τουλάχιστον ποιος θα είναι ο επικεφαλής, ποιος θα ηγείται του συνδυασμού. Μετά, αυτό είναι το επίπεδο. Το δεύτερο πρόβλημα είναι η τάση, η οποία είναι κατιούσα τα τελευταία χρόνια. Δεν είναι ε, πολύ σοβαρό πρόβλημα, αλλά αυτό είναι το περίεργο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και στις 28 χώρες μέλη υπήρχε μεγαλύτερο ποσοστό αύξηση στις εθνικές ε, εκλογές ως προς τη συμμετοχή ε, στο διάρκεια των 70 ετών που έχουμε ευρωεκλογές, αν λάβουμε υπόψη το θέμα αυτό. Από το 1979 που έχουμε ευρωεκλογέ, συγγνώμη. Δεν μπορούμε να λέμε ότι δεν λειτουργεί τίποτα, ότι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν πάνε καλά τα πράγματα και επειδή δεν πάνε καλά τα πράγματα ο κόσμος δεν ψηφίζει. Είναι πολύ απλοϊκή αυτή η νοοτροπία και νομίζω ότι ο πιο εύκολος ε, τρόπος να προχωρήσουμε, που δεν απαιτεί και αλλαγή της συνθήκης, είναι να συνεχίσουμε αυτό που ξεκινήσαμε σε αυτές τις ευρωεκλογέ, που εν μέρη είχε αποτέλεσμα, γιατί τελικώς μας οδήγησε σε έναν ε, ε, πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αν το ε, γνωστοποιήσουμε αυτό, ε, ε, το μάθει περισσότερο κοινή γνώμη και το χρησιμοποιήσουμε αυτό ως κινητήριο μοχλό θα προχωρήσει. Θα πρέπει να επικεντρωθούμε λοιπόν σε αυτό που έχει σημασία και να δούμε και ποια σημεία έχουν και λιγότερες αντιστάσεις. Ο κύριος Καζιμίρ. Ευχαριστώ πολύ. Αν δούμε τους ευρωπαϊκούς εκλογικούς νόμους, τότε νομίζω ότι δεν μπορούν και πολλοί να μεταρρυθμιστούν. Δεν είναι τομέας όπου εύκολα μπορεί να οικοδομηθεί εμπιστοσύνη προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στο κέντρο της συζήτησής μας εξετάσαμε το θέμα των πολυεθνικών ψηφοδελτίων ή τις λεγόμενες, τα λεγόμενα πανευρωπαϊκά ψηφοδέλτια. Και αυτό βέβαια πρέπει να υπάρχουν και πανευρωπαϊκά κόμματα. Είναι τελείως τεχνητή η δομή αυτό το πράγμα. Ο καθηγητής Ραντζέλ μας μίλησε για το μύθο του Σισίφου και νομίζω, ότι, νομίζω όμως ότι στην πραγματικότητα πρόκειται μάλλον για φαρσοκομωδία του Μολιέρου. Μιλάμε για έναν λαό ή δήμο που δεν υπάρχει. Και εμείς μιλάμε για έναν μη υπάρχοντα ευρωπαϊκό δήμο ή εκλογικό σώμα. Είναι τελείως τεχνητά όλα αυτά. Δεν υπάρχει ευρωπαϊκός λαός. Και κάποιος είπε σωστά ότι ούτε καν υπάρχει κοινός ευρωπαϊκός δημόσιος χώρος. Γιατί ένας Γάλλος σοσιαλιστής ψηφοφόρος να νιώσει την ανάγκη να ψηφίσει κάποιο ψηφοδέλτιο όπου θα συνυπάρχει και ένας Ιταλός ή Βρετανός σοσιαλδημοκράτης. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα και αφού δεν υπάρχει αυτός ο δημόσιος χώρος. Είναι όλα τεχνητά λοιπόν και άρα ε, είναι αδιέξοδο. Ο κύριος Ρετοντσίνη απ' την άλλη όταν μίλησε μας είπε για μεγαλύτερες, ευρύτερες πολιτικές ισοματώσεις που θα ήταν διατεθειμένες και να χάσουν τις ευρωεκλογέ. Αυτά είπε. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όμως δεν είναι χαρακτηριστικό τυπικό που κοινοβούλιο. Σπανίως στα εθνικά κοινοβούλια υπάρχουν συνασπισμοί όπως εκείνοι που δημιουργούνται στο Ευρωπαϊκό. συνασπισμοί που καλύπτουν ευρύτερο πολιτικό φάσμα από ό,τι γίνεται συνήθως στα εθνικά κοινοβούλια και θα ήταν πολύ δύσκολο νομίζω να μιλήσει κανείς για την κανονική δημοκρατική αντιπαλότητα όπως γίνεται στα κράτη-μέλη. Το καλύτερο λοιπόν, το μόνο που θα μπορούσαμε να κάνουμε αν θέλουμε να επανέλθει ή να αυξηθεί η αξιοπιστία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ήταν μερικές μικρές μεταρρυθμίσεις, ελάσσονες, αλλά με ρεαλιστική βάση, μάλλον, όπως καλύτερο έλεγχο της Κομισιόν και αυτή η συνεχιζόμενη ο συνεχιζόμενος μερικός έλεγχος της Κομισιόν από το Κοινοβούλιο δεν αρκεί πια. Δεν είναι αρκετά αυστηρός και ακριβής. Δεν είναι όπως οι έλεγχοι που κάνουν τα εθνικά κοινοβούλια για την εξουσία, εκτελεστική εξουσία. Όσο για την Ευρωπαϊκή Νομοθετική Πρωτοβουλία. Και αυτό πρέπει να μετακινηθεί πρέπει να μπορούν και οι πολίτες να έχουν κάποιο λόγο σε αυτά στη συνθήκη της Λισαβόνας δίνονται τέτοιες δυνατότητες για συζήτηση, μεταρρύθμιση, τροποποίηση της νομοθεσίας και είναι και αυτό κάτι που η πρωτοβουλία των πολιτών θα έπρεπε να απευθύνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό θα ήταν μια ενδιαφέρουσα αλλαγή που θα μπορούσαμε να κάνουμε. Και είναι τομέα όπου μπορούμε να κάνουμε μια προσπάθεια να ενδυναμώσουμε τις δυνατότητες των Ευρωπαίων πολιτών. Αλλά βέβαια αυτό σημαίνει και καλή συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκού και Εθνικών Κοινοβουλίων. Με την βάση της επικουρικότητας βέβαια θα μπορούσαμε όλα αυτά να τα δούμε βαθμιαία και προοδευτικά με βάση αυτά τα στοιχεία και τότε νομίζω θα μπορέσουμε να ενισχύσουμε την αξιοπιστία και το κύρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ενώ τα λεγόμενα πανευρωπαϊκά ψηφοδέλτια νομίζω δεν είναι ρεαλιστικά πράγματα. Διότι ακριβώς δεν υπάρχει πανευρωπαϊκή συνείδηση για την ύπαρξη ενός ευρωπαϊκού λαού. Σας ευχαριστώ πολύ. Η Mercedes Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Πρόεδρε. Καταρχάς, εγώ διαφωνώ με τον συνάδελφο Ιοντόσκι. Δεν θεωρώ ότι κάποιος ε, προσπαθεί να ε, ξεφύγει από την πραγματικότητα για τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα. Βέβαια, όποιος δεν συμμετέχει σε ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα θεωρεί ότι δεν υπάρχουν. Στην πραγματικότητα υπάρχουν και στην πλειονότητα των χωρών μελών πήραν και τις περισσότερες ψήφους. Κόμματα που είχαν μια σαφή ε, υποψηφιότητα και υποψήφιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και έχουν και ε, συγκεκριμένη ε, ταύτιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο γιατί πολλά χρόνια συμμετέχουν στο αντίστοιχο ευρωπαϊκό τους κόμμα. Αν θέλουμε λοιπόν να επικεντρωθούμε στην ουσία, θα πρέπει να επικεντρωθούμε κυρίως σε έναν ευρωπαϊκό εκλογικό νόμο, ο οποίος δεν θα ασχολείται με άλλη τα περίπου θέματα όπως το θέμα της ε, απλής αναλογικότητας. Διότι αν αρχίσουμε να μπαίνουμε στο ναι. θέμα της κατανομής των εδρών μεταξύ των χωρών μελών ή τη λίστα δεν θα καταφέρουμε τίποτα. Θεωρώ επίσης ότι το θέμα της συμμετοχής ε, στις εκλογές θα πρέπει να αξιολογηθεί με λίγο πιο πολιτικό τρόπο, διότι Όλο ένα και περισσότερο το θέμα της ε, ε, μη συμμετοχής είναι μία πολιτική ένδειξη. Βεβαίως με εκλογικούς νόμους από τους δικούς μας είναι περισσότερο μία πολιτική ένδειξη για το τι γίνεται στο εσωτερικό της χώρας και όχι στην Ευρώπη. Αλλά αυτή τη φορά, κατά την άποψή μου, υπήρχε και μία πολιτική ένδειξη προς την Ευρώπη. Δηλαδή μία επίκριση ως προς τον τρόπο με τον οποίο η Ευρώπη διαχειρίστηκε την οικονομική κρίση πιο γενική, πιο συγκεκριμένη, ε, εξαρτάται από κάθε χώρα, αλλά τελικώς αυτό είχαμε. Ιδίω αν εξετάσει κανείς τι γίνεται όταν υπάρχουν σκάνδαλα, προβλήματα, ε, το γεγονό ότι ο κόσμο δεν αποδέχεται τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώστηκαν τα σοβαρά προβλήματα, κυρίω η ευρωπαϊκή οικονομία. Εκεί όχι μόνο αλλάζουν οι συσχετισμοί των ψήφων, αλλά αλλάζει και η συμμετοχή σε ευρωεκλογέ ω ένδειξη ότι δεν θέλω να αλλάξω κόμμα, γιατί πιστεύω τα ίδια πράγματα, αλλά δεν θέλω να αποδεχτώ ω σωστά αυτά τα οποία έκαναν όλοι. Και αυτό θεωρώ ότι είναι μια πολύ σημαντική ένδειξη που νομίζω ότι την αντιλήφθηκε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία πρότεινε να αλλάξουμε στάση και άρχισε να μιλάει και πάλι για να, επενδύσεις, ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων απασχόληση. Θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει κυρίως να προσπαθήσουμε να δώσουμε μεγαλύτερη νομιμοποίηση στον Ευρωπαϊκό Εκλογικό Νόμο, να μην επισέλθουμε σε θέματα κατανομής εδρών μεταξύ των χωρών. Εγώ θεωρώ ότι η αρχή που προτείνεται από τον καθηγητή ε, Πούκελσχάιμ για την πιθανή διπλή αναλογικότητα, ακόμα και αν ε, παρουσιάζει κάποια προβλήματα, ε, μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε και είναι ενδιαφέρουσα διότι μας επιτρέπει αυτή τη δυνατότητα να έχουμε μια διτή σύνδεση με τον αριθμό των ευρωβουλευτών που εκλέγονται σε κάθε χώρα, αλλά ταυτόχρονα και με τα αποτελέσματα και τις εκλογικές πολιτικές. Τα πολιτικά και εκλογικά αποτελέσματα είναι πάρα πολύ σημαντικά, διότι ε, από την ε, ιδέα του speech and candidate δεν υπάρχει επιστροφή, δηλαδή το γεγονός ότι τα μεγάλα κόμματα θα έχουν πάντα έναν υποψήφιο για πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα ψηφοδέλτια τους. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε ώστε να δημιουργήσουμε έναν εκλογικό νόμο ε, στην οποία η συμμετοχή σε μια ευρωπαϊκή εκλογική παράταξη που έχει την αντίστοιχη ιδεολογία με το Εθνικό ε, Κόμμα είναι ένα και πιο σημαντικό στοιχείο. Εγώ προσωπικώς έχω μία πρόταση αντίστοιχη με αυτή του καθηγητή Πούκελσχάιμ. Αντί να προσθέσουμε ε, ένα πανευρωπαϊκό ψηφοδέλτιο, μια πανευρωπαϊκή λίστα, να υπάρχει η υποχρέωση να συμμετέχει κάποιο σε ένα ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα προκειμένου να μπορεί να είναι υποψήφιος σε ευρωεκλογέ. Δεν μπορεί να είναι το θέμα των ορίων το πρόβλημα ε, για μένα δεν χρειάζεται να υπάρχει όρια, διότι το όριο θα μπορούσε να λύνεται από το γεγονός ότι θα πρέπει να υπάρχει συμμετοχή σε ένα ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα που να έχει μια ελάχιστη εκπροσώπηση στην Ευρώπη. 8-10 χώρες παραδείγματος χάρη. Αναφερόμαστε σε ευρωεκλογέ, η νομιμοποίηση απορρέει από την εκπροσώπηση ε, από ένα πολιτικό κόμμα ευρωπαϊκό και από το γεγονός ότι αυτό το κόμμα ανταποκρίνεται στους κανόνες της δημοκρατικότητας των κομμάτων όπως καθορίζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό θα μας επέτρεπε να μην πρέπει απαραίτητος να σκεφτούμε ε, μια πανευρωπαϊκή λίστα, αλλά να υπάρχει μια εγγύηση ότι όλοι οι αιρετοί θα προέρχονται από συνασπισμούς ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και αυτοί οι συνασπισμοί θα εκπροσωπούν το σύνολο των Ευρωπαίων πολιτών και όχι ο καθένας ε, το εθνικό του κόμμα. Επίσης, εγώ είμαι πεπισμένη ότι και η πλειονότητα των Ευρωπαίων πολιτών αρχίζει να έχει μια πολιτική συνάφεια με την ευρωπαϊκή πολιτική. Ακόμα βέβαια είναι διπλή αυτή η συνάφεια, αλλά αυτό είναι δεδομένο. Είναι σαν τη διπλή υπηκότητα. Εμείς νιώθουμε ε, πολίτες της χώρας μας και πολίτες της Ευρώπης, τουλάχιστον αυτοί που είναι υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και το ίδιο αυτό, εγώ νιώθω ότι είμαι τμήμα του Ιταλικού πολιτικού μου κόμματος, αλλά ότι είμαι και τμήμα του Ευρωπαϊκού μου πολιτικού κόμματος. Είναι σαφές ότι ε, αν βαθμιδών οι προεκλογικές εκστρατείες δημιουργηθούν με το σύμβολο του Ευρωπαϊκού Πολιτικού Κόμματος το οποίο συμμετέχει το Εθνικό Κόμμα, αυτή η έννοια της συνάφειας με το κόμμα θα αυξάνονταν. Και ε, το γεγονός ότι θα νιώθει κάποιος ότι ανήκει σε μια ευρωπαϊκή πολιτική οικογένεια μπορεί να έχει και ε, ε, συνέπειες για την πολιτική μάχη στην Ευρώπη. Δεν χρειάζονται μεγάλες ε, εκστρατείες επικοινωνίας, χρειάζεται να υπάρχει και αυτή η αίσθηση της πολιτικής μάχης και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να είναι σαφές ότι αυτό θα μας οδηγήσει σε ένα πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θεωρώ ότι θα πρέπει να δούμε και κάποιε από τις προτάσεις του κυρίου Μπερτοντσίνη, κυρίως ε, ως προς το γεγονός ότι αν και συνήθως θα πρόκειται για συνασπισμούς, για προφανείς λόγους, ε, λόγω της ε, πολυπλοκότητας της Ευρώπης, 28 χώρες, πολύ διαφορετικές πλειοψηφίες σε κάθε χώρα, αλλά να υπάρχει τουλάχιστον η δυνατότητα, ακόμα και μέσω εκλογικών μηχανισμών, ε, αν όχι να γίνεται αναλλαγή, να υπάρχει τουλάχιστον μια ευελιξία. Να μην είναι δε και καλά πάντα ο ίδιος συνασπισμός ο οποίος λόγω του εκλογικού μηχανισμού θα ε, κάνει υποχρεωτική αυτή τη συμφωνία να υπάρχουν κάποιες διακυμάνσεις και κάποιες αλλαγές σε κάποιο βαθμό. Θεωρώ ότι θα ήταν χρήσιμο επίσης να εξετάσουμε και το γεγονός ότι τα πολιτικά κόμματα τα οποία ε, παρουσιάζονται ως συνασπισμός ε, στις ευρωεκλογέ να μην έχουν μόνο ένα σύμβολο, να έχουν και ε, κάπου ένα πρόγραμμα. Δεν χρειάζεται να είναι τόμο αυτό, μπορεί να είναι ένα φυλάδιο με ένα πρόγραμμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μπορούν να προσθέσουν και σε εθνικό επίπεδο κάποια πράγματα, αλλά να φαίνεται σαφώ ποια είναι η πολιτική πρόκληση των ευρωεκλογών και επομένω ποια πράγματα θα προτείνει να κάνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο το συγκεκριμένο πολιτικό κόμμα. Και βεβαίω αν το επιθυμούν μπορούν στην ίδια λίστα να υποδεικνύουν και τον υποψήφιο πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αυτούς. Αυτό σημαίνει ότι αναλαμβάνουν πλήρως την ευθύνη ενώπιον των πολιτών του ευρωπαϊκού τους ρόλου και όχι μόνο του εθνικού τους ρόλου. Εγώ θεωρώ ότι θα έπρεπε να επεξεργαστούμε αυτά και να μην δούμε τα θέματα της εκπροσώπησης της κάθε χώρας, διότι η τροποποίηση ε, της κατανομής των εδρών ε, στο Κοινοβούλιο σαφέστατα θα πρέπει να συνοδεύεται και από αντίστοιχη τροποποίηση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Νομίζω δεν έχουν οριμάσει ακόμα οι συνθήκες γι' αυτό και θα ξεκινήσουν μάχες για να προασπίσει ο καθένας τις δικές του εθνικές έδρες και δεν νομίζω ότι χρειάζονται αυτές οι μάχες διότι υπάρχει η αρχή της αναλογικότητας και η αρχή της φθήνουσας αναλογικότητας δεν ε, αλλάζει λόγω των, ε, του μεγέθους των πολιτών των ευρωπαϊκών χωρών. Ίσως θα μπορούσαν να γίνουν κάποιες μικρές αλλαγές αν ε, καταλήξουμε σε κάποια συμφωνία για την ένταξη μιας νέας χώρας θα μπορούσε ίσως επί τη ευκαιρία να γίνει και κάποια μικροαλλαγή. Αλλά δεν νομίζω ότι θα καταφέρουμε να προχωρήσουμε πολύ ε, περαιτέρω και δεν νομίζω ότι είναι και στις βασικές μας απαιτήσεις. Το να υπάρχει μεγαλύτερη εκπροσώπηση των μικρών ε, είναι μία ανάγκη στον τρόπο με τον οποίο δημιουργήθηκε η Ευρώπη και νομίζω ότι θα συνεχίσει να οικοδομείται και κατά αυτόν τον τρόπο. Να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές, διότι βρήκα πολύ ενδιαφέρουσες τις παρεμβάσεις και μας έδωσαν πάρα πολλά στοιχεία για να συζητήσουμε. Ευχαριστώ. Πέντρο Σίλβα Περέιρα στη συνέχεια και θα ζητήσω από τους εμπειρογνώμονες να λάβουν το λόγο μετά. Um Ευχαριστώ. Πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Πρέπει όμως να μην ξεχάσουμε, δεν πρέπει να ξεχάσουμε ότι η συζήτηση γίνεται σε ζωτική εποχή για την Ένωση, σε κρίσιμη εποχή. Εποχή απογοήτευσης των πολιτών από τα αποτελέσματα της δράσης των ευρωπαϊκών θεσμών και εποχή όπου οι πολίτες αμφισβητούν την νομιμότητα των αποφάσεων που παίρνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και το θέμα γίνεται όλο και σοβαρότερο καθώς οι αποφάσεις μας αφορούν όλο και περισσότερο τα χρηματικά και τον προϋπολογισμό και τα δημοσιονομικά. Είναι λοιπόν βασικό να ενδυναμωθεί η αναλογικότητα και μάλιστα η διπλήτη αυτή. Δεν πρέπει η αγνή και άδολη αναλογική να μην συνοδεύεται με κάτι ανάλογο και στο Συμβούλιο για να υπάρχει ισότητα αλλιώς. Θα χειροτερέψει το αίσθημα που έχουν πολλοί πολίτες, ιδιαίτερα σε μικρομεσαίου μεγέθους κράτη. Για αυτές τις χώρες θα ήταν απαράδεκτη χειροτέρεψη του δημοκρατικού ελλείμματος και στο χειρότερο μάλιστα χρονικό σημείο. Δεν γίνονται αυτά. Δεύτερον, πρέπει να δούμε το θέμα της αποχής. Δεν είναι πρόβλημα που οφείλεται στο εκλογικό σύστημα το ίδιο. Αυτό το έχουν πει και άλλοι ούτε είναι κάτι που καμένα μπορεί να λυθεί με υποχρεωτική ψήφο όπως δεν μπορεί να λυθεί και με τεχνητές λύσεις όπως είπε και ο Ρομπέρτο Νταλιμόντε. Οφείλεται κυρίως στο αίσθημα ότι οι ευρωεκλογέ δεν παίζουν κανέναν αποφασιστικό ρόλο. Αυτό όμως σημαίνει ότι το χειρότερο που θα μπορούσε να γίνει θα ήταν να υπαναχωρήσουμε εμείς, δηλαδή να χωρίσουμε τις ευρωεκλογές να γίνονται οι ευρωεκλογέ την ίδια στιγμή με τις εθνικές αυτό θα ήταν ό,τι χειρότερο θα μπορούσαμε να κάνουμε θα αυξανόταν η συμμετοχή βέβαια αλλά θα επανεθνικοποιούσε τις ευρωεκλογέ και θα έπαβε πια να ισχύει οποιαδήποτε έννοια αποφασιστική σημαντικής εκλογικής διαδικασίας για τα ευρωπαϊκά. Και τέλος, κάτι που νομίζω ότι έχει σημασία και που πρέπει να το πετύχουμε είναι ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες πρέπει να καταλάβουν το ρόλο που μπορούν να παίξουν οι ευρωεκλογέ και άρα να αυξηθεί η ορατότητα της ευρωπαϊκής πολιτικής ζωής. Να τονίσουμε τη σύνδεση που υπάρχει μεταξύ της ψήφου των πολιτών και της κατεύθυνσης που θα ακολουθεί η Ευρώπη. Έχουν ακουστεί πολλές ιδέες όπως να πρέπει ο Spitzenkandidat να αναφέρεται ρητά στα ψηφοδέλτια και οι πολιτικές, τα σύμβολα των πολιτικών ομάδων, τα σήματα να αναφέρονται στα ψηφοδέλτια και αυτό θα αύξανε νομίζω την ορατότητα και θα ήταν μέτρο σωστό. Δεν θα έλυνε άμεσα το πρόβλημα, αλλά δεν μπορεί να λυθεί άμεσα με καμία νομοθετική αλλαγή ή με άλλον τεχνητό τρόπο. Ευχαριστώ. If you could accept to speak now in the... Μήπως μπορείτε να δεχτείτε τώρα να απαντήσετε με την αντίθετη σειρά. Ναι, ναι, ναι. Σύντομα. η προοδευτική αναλογικότητα. Εστιάζεται στην ισορροπία μεταξύ πολιτικών δυνάμεων, όχι κρατών μελών. Εγώ δεν προτείνω καμία αλλαγή στην κατανομή εδρών μεταξύ κρατών μελών. Απλά υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις και λογικό είναι όταν αλλάζουμε την ε, εκλογική περιφέρεια, αν γίνει κάπως πιο μακροπεριφερειακή ή εάν χρησιμοποιήσουμε τη δυνατότητα 2 ορίου 3-4-5% αυτό σημαίνει πως μόνο οι μεγάλες πολιτικές δυνάμεις θα εκπροσωπούνται στο ε, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, όταν λέω μεγάλη εννοώ 3-4-5% έτσι δεν είναι μόνο τα μεγάλα κόμματα και μετά το άλλο. Αυτό το οποίο απαιτείται είναι ε, να πάμε, ε, να κινηθούμε σε αυτές τις γραμμές ε, στα μεγαλύτερα κράτη-μέλη. Αν δούμε το πώς χρησιμοποιούνται τα όρια ή αν δούμε τα κράτη-μέλη στα οποία υπάρχουν μάκρο περιφερειακές εκλογικές περιφέρειες βλέπουμε πως κάποια κάτι μέλη ακόμα δεν επηρεάζονται. Οπότε ίσως θα μπορούσαμε να δούμε χώρες όπως Ισπανία, Ρουμανία, Ελλάδα, Τσεχία ε, είτε υποχρεωτικά είτε προωθώντας βέλτιστες πρακτικές με γενικό στόχο περισσότερη σαφήνεια στις ευρωεκλογές ή μετά τις ευρωεκλογές. Δηλαδή, ναι, πιο σημαντικές πολιτικές δυνάμεις, πολλές πολιτικές ομάδες ακόμα, αλλά σε τελική ανάλυση μια δυνατότητα για σαφείς συνασπισμούς με μια ποικιλόμορφη βάση, όπως είπε η κυρία Μερσέντες Πέσο. Ο κύριος Ολύρη έφυγε, δεν ήξερα ότι έπρεπε να φύγει, λοιπόν, ο καθηγητής Νταλιμόντε. Χωρίς μικρόφωνο. Can you hear me now? Yes. I like to... Θα ήθελα να τονίσω αυτό το οποίο είπα και πριν. Θεωρώ πως αυτό το οποίο έκανε το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο για την εναρμόνιση των 28 εκλογικών συστήματων είναι θετικό κατά την άποψή μου είναι πάρα πολύ δύσκολο να πάμε παραπέρα από αυτό. Γιατί, τι μπορεί να αλλάξει για ένα πιο ομοιόμορφο εκλογικό σύστημα, δεν έχει τόσο σημασία. Αυτό το οποίο μετράει ε, δεν μπορεί να αλλάξει από την άλλη. Οπότε αυτή τη στιγμή το ε, Κοινοβούλιο έχει φτάσει σε μια θέση ισορροπίας. μεγαλύτερη αλλαγή, μεγαλύτερη αδύναμη αλλαγή είναι το όριο. Αλλά είναι αδύνατο νομίζω να βρεθεί μια συμφωνία μεταξύ 28 κρατών για ένα ενιαίο όριο. Και επειδή το μέγεθος των εκλογικών περιφερειών δεν μπορεί να αλλάξει, οι υπόλοιπες αλλαγές μετά δεν έχουν σημασία. Οπότε τονίζω το ότι ε, ε, αυτό είναι, έχουμε ένα σημείο ισορροπίας. Αλλά και πάλι θα πρέπει οι βουλευτές και το Κοινοβούλιο να απαντήσουν το ερώτημα. Όχι για μένα, για τον Ευρωπαίο πολίτη. Γιατί χρειαζόμαστε ομοιόμορφη εκλογική διαδικασία. Ποιος ο στόχος ο στόχος είναι να αυξηθεί η αναλογικότητα. Αν ο στόχος είναι να αυξηθεί η αναλογικότητα, επανερχόμαστε σε αυτό το οποίο είπα. Πως είναι πάρα πολύ δύσκολο να αλλάξει το όριο και αδύνατον να αλλάξει το μέγεθος των εκλογικών περιφερειών. Οπότε και αυτός ο στόχος ακόμα επιθυμητός ή όχι, γιατί μπορεί να διαφέρουν οι απόψει. κατά την απόψη μου δεν είναι επιθυμητό. μπορεί να είναι επιθυμητό για άλλου. αλλά ακόμα και αυτός ο στόχος ε, δεν μπορεί να επιτευχθεί. Το τελευταίο μου σχόλιο. Εγώ είπα πως ε, αυτά τα οποία είπα για το εκλογικό σύστημα ήταν ευσεβή πόθη. Όχι μόνο γιατί θεωρώ πως δεν υπάρχει συνένεση επί των προτάσεων DAF. Ακόμα λιγότερη συνένεση θα υπάρχει για την πρόταση Νταλιμόντε για ένα μπόνους εδρών. Αλλά για να επανέλθω σε αυτό το οποίο είπε ο συνάδελφος εδώ ο κύριος Μπερτοντσίνη. Θέλουμε πραγματικά αποφασιστικές, αποφασιστικότητα των εκλογών. Εντάξει, για τη χώρα μου ε, εμένα μου αρέσει, αλλά στην περίπτωση ε, του κοινοβουλίου αυτού κάτι τέτοιο θα σήμερα να έχουμε ένα εκλογικό σύστημα το οποίο θα προωθούσε εναλλαγή εξουσίαν, εξουσίας. Ένα ευρωπαϊκό σύστημα κομμάτων που θα επέτρεπε και θα προωθούσε αυτήν την αλλαγή. Στα χαρτιά μοιάζει μια καλή ιδέα κάτι τέτοιο γιατί θα δώσει την ευκαιρία στους Ευρωπαίους ψηφοφόρους να εκφραστούν με το να διώξουν την κυβέρνηση και να καταστήσουν την αντιπολίτευση. Μια τέτοια αλλαγή και δημοκρατική λογοδοσία μπορεί να σταματήσει την ορμή των αντιευρωπαϊκών κομμάτων. Όμως, μπορεί το κοινοβούλιο αυτό να λειτουργήσει με ένα τέτοιο μοντέλο τέλειου ανταγωνισμού. Δεν είμαι σίγουρος. Δεν είμαι σίγουρος για το εάν είναι αυτό το σωστό είδος ανταγωνισμού και σχηματισμού κυβερνήσεως. Αυτό το ανταγωνιστικό σύστημα ή εάν το σύστημα αυτό λόγω της φύσης της Ένωσης πως θα ήταν καλύτερο να έχει ένα ελβετικό μοντέλο, ένα μοντέλο συνενετικό ή το παλιό ολλανδικό μοντέλο των παράλληλων πυλώνων της κοινωνίας. Δεν ξέρω, εσάς περιμένω να ακούσω. Κύριος Πούκελσάιν. Θα ήθελα να απαντήσω με κάποιες ε, παρατηρήσεις, ε, μια χούφτα παρατηρήσεις, οπότε πέντε δάχτυλα έχω, πέντε σημεία θα πω. Λοιπόν, το πρώτο είναι ο ρόλος μας, ο ρόλος ο δικός μας. Εμείς ως μαθηματικοί δεν προτείνουμε ένα σύστημα. Και το είπα στην εισαγωγή μου, πως βασιζόμαστε στα έγγραφα της Επιτροπής σας και του Κοινοβουλίου και προσπαθούμε να δούμε τους δικούς σας πολιτικούς στόχους και ε, μετά να δούμε αν συμφωνούν με μια διαδικασία ασφαλή γιατί μοιραία οι εκλογές στο τέλος έχουν νούμερα καταμέτρηση των ψήφων και τις έδρες που καταλαμβάνεται πάλι αριθμούς δηλαδή και Βεβαίω ε, τα αριθμητικά στοιχεία πρέπει να πηγαίνουν παράλληλα με τους δικούς σας τους πολιτικούς στόχους. Βεβαίω, ε, ως μαθηματικός ε, και καθηγητής έχω τη φιλοδοξία ο κόσμος να καταλαβαίνουν το σύστημα. Ο βουλευτής ο κύριος Βίλαντ είπε πως θέλει τα τρία τέταρτα των δασκάλων και των καθηγητών να μπορούν να το καταλαβαίνουν. Εγώ θα ήθελα να το καταλαβαίνουν και 100% των βουλευτών. Να καταλαβαίνετε το σύστημα με το οποίο εκλέγεστε δηλαδή. Δεύτερον, προσπάθησα να εξηγήσω την διπλή αναλογικότητα και θα ήθελα και πάλι να πω πως είναι το βασικό μας ε, μήνυμα σήμερα. Η διπλή αναλογικότητα μας επιτρέπει να αποσυνδέσουμε το πρόβλημα της εκπροσώπησης του κράτους μέλους από το πρόβλημα της ε, πολιτικής ε, διαίρεσης του εκλογικού σώματος. Η γραπτή μας δήλωση ήταν δομημένη με βάση αυτά τα οποία έλεγε ε, η κυρία Χίμπνερ στην πρόσκλησή της ε, όπου δεν γινόταν λόγος για την ε, σύνθεση από πλευράς εθνικών αντιπροσωπιών. Και... Και βέβαια υπάρχουν αυτά τα δύο επίπεδα, η πολιτική διαίρεση και η εδαφική κατανομή του εκλογικού σώματος. Η πολιτική κατανομή ε, ήταν εκεί που δώσαμε βάρος. Με αυτό ακριβώς ζήτησα ε, ισότητα της ψήφου. Εγώ όταν βλέπω το ψηφοδέλτιο δεν ε, σημειώνω το αν είμαι Γερμανός ή Πορτογάλος ή Ιταλός, ψηφίζω ένα κόμμα. Και το ερώτημά μου, το ερώτημά μας σε εσά ως Επιτροπή είναι θέλουμε πολιτική ισότητα όταν ψηφίζω εγώ ένα κόμμα και βάζω το σταυρό και κάποιος άλλος στη Μάλτα ψηφίζει το ίδιο κόμμα και στην Ιρλανδία μετράει το ίδιο η ψήφος μας όσον αφορά το τελικό αποτέλεσμα. Αυτό σημαίνει η ισότητα της ε, ψήφου. Το ότι δεν υπάρχει αυτό συνθήκες κατά την απόψή μου είναι νομίζω πως αυτή η φθήνουσα αναλογικότητα βεβαίως δεν ικανοποιεί τον ψηφοφόρο. Και βέβαια υπάρχει και η δεύτερη αυτή διάσταση την οποία αναφέρεται, την οποία μπορούμε να τη δούμε ανεξαρτήτως. Το τέταρτο σημείο ε, είναι ως απάντηση στον κύριο Λάινεν, γιατί καταλήξαμε σε πανευρωπαϊκά κόμματα εσείς ε, θα αποφασίσετε ποια κόμματα θα ε, κατέβουν στις εκλογές. Ε, απλά βασιστήκαμε στο ότι ο τωρινός ε, ορισμός του Ευρωπαϊκού Κόμματος είναι περιοριστικός και είναι κατανοητό γιατί θέλετε να χρηματοδοτήσετε κάτι το οποίο θα έχει ήδη κάποια ουσία. Αλλά βεβαίως επαφίεται τελικά στους ψηφοφόρους, στους εκλογείς και Εμεί θεωρούμε πω θα πρέπει να είναι πιο ανοιχτό, φιλελεύθερο ο ορισμό και όχι τόσο περιοριστικό. Αλλά εμεί είμαστε, όπω είπα, μαθηματικοί. Εσεί θα τα διατυπώσετε. Πέμπτον, η διπλή αναλογικότητα απαιτεί πανευρωπαϊκά κόμματα ή κόμματα στο ευρωπαϊκό επίπεδο ή όπως θέλετε πείτε το. Τώρα ε, τίθεται το ζήτημα η κότα έκανε το αυγό ή το αυγό την κότα. Θέλουμε δηλαδή τα ευρωπαϊκά κόμματα να κατεβαίνουν στις εκλογές και να φαίνονται με πρόγραμμα επιθυμητό, αλλά το αν θα προκύψει τόσο γρήγορα δεν ξέρω. Αυτό το οποίο μπορώ να πω είναι πως όταν μιλάμε για τα νούμερα, ο ρόλος των ευρωπαϊκών κομμάτων είναι πολύ αδυναμός. Δηλαδή απλά λειτουργούν ως ένας τρόπος να κάνουμε ένα άθροισμα. Λέμε ότι ανήκω σε αυτή την οικογένεια και μετά θρίζουμε τις ε, ψήφους και υπολογίζουμε και βγάζουμε το νούμερο. Οπότε ε, πρόκειται για μια πάρα πολύ ασθενική λειτουργία των ευρωπαϊκών κομμάτων αν απλά χρησιμεύουν για να κάνουμε το άθροισμα των εθνικών. Αλλά θα μπορούσαμε νομίζω να ε, πάμε σε μια διπλή αναλογικότητα και επανερχόμαστε στο αυγό και την κότα όταν ξεκινήσουν να λειτουργούν έτσι θα ε, κατεβαίνουν και στις εκλογές με πολιτικούς όρους. Ευχαριστώ, Um, Νομίζω ότι αυτή είναι η κοστή τέτοια συζήτηση που έχω κάνει στο Κοινοβούλιο εδώ για τα θέματα αυτά. Και κάθε φορά ε, εμπλουτίζεται και γίνεται πιο ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Θα ήθελα καταρχάς να τονίσω ότι εμείς δεν αναζητούμε ομοιομορφία έτσι για την ομοιομορφία δεν είναι μια ε, ακαδημιακή διαδικασία. Η αναζήτηση δημιουργίας ενός Ομοσπονδιακού Κοινοβουλίου που ζητά την εμπιστοσύνη του εκλογικού σώματος. Είναι αυτό. Εγώ δεν ενδιαφέρομαι να ορίσω τι είναι δήμος ε, και δημόσιος χώρος. αλλά θέλω το Κοινοβούλιο να γίνει το μόνο πολιτικό βήμα της ενιαίας πολιτικής αγοράς. Εδώ θα αποφασίζεται, όχι αποκλειστικά, αλλά σε εταιρική σύμπραξη με την άλλη Βουλή. Εδώ είναι ο χώρος στον οποίο λοιπόν θα αποφασίζεται το μέλλον της Ευρώπης. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι ιστορικά σημαντικό, είναι πάρα πολύ σημαντικό τη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία που είναι κομβική σημασίας και η δημοκρατική κοινωνία είναι η πιο ευάλωτη από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας μεγάλος συμβιβασμός μεταξύ της Διεθνούς Αρχής Δικαίου της Ισότητας των Κρατών αφενός και της Δημοκρατικής Αρχής του ένας άνθρωπος μία ψήφος. Και ο καθορισμός του συμβιβασμού είναι αυτός ο οποίος θα μας επιτρέψει να βελτιώσουμε την ποιότητα και την ισχύ της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας. Δεν υπάρχει τέλειο σύστημα, όπως ε, συνεχώς καταδεικνύουν οι συζητήσεις εδώ, αλλά αυτό που έχει σημασία θεωρώ είναι οι διαδικασίες και οι κανόνες ε, που αφορούν τα θέματα αυτά να γίνουν πιο μεθοδικοί και να μην είναι αυθαίρετοι όπως είναι τώρα. Εγώ δεν θεωρώ ότι η διαπραγμάτευση για τις έδρες μεταξύ των κρατών μελών νωρί το πρωί ή στο τέλος κάθε διακυβερνητικής συνδιάσκεψης είναι υπεύθυνο τρόπος να κάνει κανείς τη δουλειά του. Δεν θεωρώ ότι αυτό σέβεται το εκλογικό σώμα με τόσο αποτελεσματικό τρόπο. Αναζητούμε λοιπόν καλύτερη μεθοδικότητα, να υπάρχει μεγαλύτερος βαθμός δημοκρατικής εμπιστοσύνης, αλλά επίσης να υπάρχει και συμμόρφωση με καθολικές αρχές συνταγματικού δικαίου. Και μπορεί να γίνει αυτό. Τίποτα δεν είναι αδύνατο. Αυτό που είναι ίσως ε, περίεργο και απίθανο και μάλλον δεν είναι λογικό είναι να συζητεί, ε, συζητά κάποιος για τα κοινοβούλια χωρίς να συζητά ε, και την κυβέρνηση και η απουσία μιας ισχυρότερης θέσης εκτελεστικής αρχής που έχει τη διακυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που οδηγεί από μόνο του στη συζήτηση ε, για τον εκλογικό νόμο και μάλιστα σε μια περίεργη συζήτηση. Γι' αυτό είπα ότι θα πρέπει οι προεκλογικέ εκστρατείε να είναι πιο η σημασία, να ενισχύσουμε την αίσθηση του επιλο... της επιλογής του ψηφοφόρου και να κάνουμε λίγο πιο δραματικές, αν θέλετε, τις διαφορές μεταξύ των πολιτικών κομμάτων και τις εντάσεις μεταξύ ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Ευρωπαϊκών Πολιτικών Κομμάτων που παρά τα προβλήματά τους αναδύονται σιγά-σιγά και τα εθνικά κοινοβούλια και τα εθνικά κόμματα που πλέον έχουν περάσει σε ένα άλλο στάδιο. Η κλίμακα και η πολυπλοκότητα των θεμάτων που συζητούμε εμείς εδώ στο κοινοβούλιο μας ε, ε, κάθε μέρα έχουν υπερκεράσει τις δυνατότητες ε, των παλιών κρατών εθνών να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα και να συμβασίζονται στις παλιές περιγραφές κρατών εθνών ε, για τη δημοκρατία. Και το να βασιζόμαστε σε αυτές τις παλιές περιγραφές ε, είναι κάτι το οποίο ε, είναι μάλλον επικίνδυνο. Ολοκληρώνω λοιπόν όπως ξεκίνησα. Θεωρώ ότι το πιο σημαντικό είναι να υπάρχει μία υπερεθνική λίστα για μία πανευρωπαϊκή έδρα για τις εκλογές του 2019. Και ο λόγος είναι κυρίως για να δημιουργήσουμε τα ομοσπονδιακά πολιτικά κόμματα και να προσπαθήσουμε να δράσουμε ως ένα δημοκρατικό σώμα το οποίο θα δράει υπέρ των πολιτών και των εθνικών ομοσπονδιακών αρχών εδώ στις Βρυξέλλες. Και για τους ε, πρώους συναδέλφους ε, εδώ στην Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων, θα ήθελα να πω πραγματικά προσπαθήστε να είστε πιο τολμηροί εδώ στην αρχή της ε, θητείας σας. Τίποτα δεν είναι αδύνατο. μπορούμε να έχουμε μια συνταγματική συνθήκη και αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν καταφέρει να δράξει αυτή την ευκαιρία, κατά πάσα πιθανότητα θα το καταδικάσει η κοινή γνώμη για πολλές γενιές ακόμα. Ευχαριστώ Άντριου. Θα ήθελα απλώς ε, να ολοκληρώσω τώρα εδώ, να κλείσουμε τη σημερινή συνεδρίαση, να ευχαριστήσω και πάλι όλους ε, και τους ομιλητές και όλους εσάς και θα επανέλθουμε στα πλαίσια της, των εργασιών μας για την έκθεση και στις προτάσεις σας. Ευχαριστώ πολύ.